Dear colleagues, uh, welcome to this um, hearing on the rule of law. Ο Πρόεδρος, γεια σας συνάδελφοι. Έχουμε τώρα την ε, παρουσίαση των αποτελεσμάτων γίνεται της ε, αποστολής στην Πολωνία, αλλά τώρα έχουμε αυτή την ακρόαση που αφορά την κατάσταση για το κράτο δικαίου στην Πολωνία, για την ανεξαρτησία τη δικαιοσύνη πιο συγκεκριμένα. Οπότε, ένα θερμό καλώ όρισε. Ε, το έχουμε οργανώσει στη συνέχεια της αποστολής μας στη Βαρσοβία για την κατάσταση του κράτους δικαίου. Αυτό έγινε στις 19 μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου του 2018. Ε, είχα την τιμή να προεδρεύσω σε εκείνη την αποστολή και το πρόγραμμα αποφασίστηκε από τις πολιτικές ομάδες. Διορθώνεται ως εξής εις τρία τμήματα από τα πρώτα Πρώτα πρώτα έχουμε τον πρώτο αντιπρόεδρο Φραντς Τίμερμανς και δυστυχώς Όσον αφορά εκπροσώπηση της Πολωνίας, καλέσαμε τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Δυστυχώς, θα πρέπει να εκφράσω την δυσόσχειά μου, διότι η κυβέρνηση δεν απεδέχθη την πρόσκλησή μας. Και σα θυμίζω, στα πλαίσια εκείνη της αποστολής μας που έγινε, όπω ανέφερα τον Σεπτέμβριο, Ούτε τότε μπορέσαμε να συνθούμε με τον Υπουργό Δικαιοσύνη για να συζητήσουμε τα των μεταρρυθμίσεων. Το συζητήσαμε πάντως με τον πρέσβη της χώρας και καταβάλαμε πάσα δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε να προσκληθεί εκπρόσωπος της κυβερνήσεως. Επίσης, η Αυστριακή Προεδρία αλλά και οι επόμενοι, οι Ρουμάνικοι, θα προβούν σε μία σύντομη δήλωση ε, σε σχέση με το άρθρο 7 παράγραφος 1. Μετά θα έχουμε εκπροσώπους της Επιτροπής της Βενετίας. Από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο ε, Δικαστικών και ε, τον Πολωνών Διαμεσολαβητή. Μετά έχουμε εκπροσώπου του μολύντων και πανεπιστημιακούς και στο τέλος θα έχουμε απαντήσει. Πριν αρχίσουμε πάντω την άκροασή ε, ε, μας, θα έχουμε παρουσίαση κάποιων συμπερασμάτων από την ε, αποστολή μας του Σεπτεμβρίου. Η έκθεση σχετική συντάχθηκε σε συνεργασία με τις πολιτικές ομάδες, με τα μέλη της αποστολής. Πρόκειται να δημοσιεύσουμε την έκθεση αυτή για την αποστολή και θα συζητηθεί αρχές του, επομένου μηνός. Θα υπάρχει και μετάφραση στα πολωνικά. Θέλαμε με την αποστολή να δούμε τι γίνεται με το σύστημα της δικαιοσύνης στην χώρα, τι κάνουν σχετικά οι αρχές της χώρας, πώς έχει η κατάσταση και αυτά στα πλαίσια ε, της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου και βέβαια εδώ σας παραμένω στο άρθρο 7 όπως το ενεργοποίησε αυτό και την ε, διαδικασία του Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύνθεμα με εκπροσώπους από την Βουλή, το Κοινοβούλιο, την Κυβέρνηση, ε, εκπροσώπους του ΑΣΕ, νομικούς, δημοσιογράφους, εκπροσώπους της κοινωνίας και θέλουμε όλους τους συνομιλητές μας να τους ε, ευχαριστήσουμε. Σας ευχαριστούμε για το χρόνο τους και για όλα όσα μας εξήγησαν. Κάνουμε κάθε προσπάθεια να συντήσουμε όσο περισσότερα μέλη της κυβέρνησης γινόταν και δυστυχώς ε, πάρα πολλές από ε, τις προσπαθειές μας συνάντησαν κλειστές πόρτες. ως πρόεδρος της αντιπροσωπείας του Κοινοβουλίου εμένω στο ότι αυτό το οποίο είναι θεμητό είναι να κάνουν οι αρχές, να κάνει η κυβέρνηση μια εκβάθρον μεταρρύθμιση στη δικαιοσύνη. Και άκουσα πάρα πολύ είχαν να πούν. Σας υπενθυμίζω τα της ιστορικής προς Ευρωπαϊκή Ένωση της χώρας και το ότι οι Πολωνοί δικαστές ενεργούν και ως Ευρωπαίοι δικαστές. Είναι καθήκον τους να ενεργούν αμερόληπτα και να εφαρμόζουν επίσης αμερόληπτα το κοινωτικό δίκαιο. Και μας προβληματίζουν όλα αυτά που έχουν γίνει μέσω αυτών των προανφερθησών μεταρρυθμίσεων και όλα αυτά οδηγούν σε μια επιρροή τη κυβέρνηση όσον αφορά τη σύνθεση, τη λειτουργία του Συνταγματικού Δικαστηρίου, των τακτικών δικαστηρίων του Εθνικού Συμβουλίου Δικαστών και το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας. Ε, οπότε με προβληματίζει το ότι το κράτος δικαίου έχει φυγεί εδώ. και ότι επίσης έχουν καταπατηθεί, υπάρχει κίνδυνος να καταπατηθούν βασικές αρχές όπως η διαίρεση των εξουσιών, η νομιμότητα, η νομική ασφάλεια, η ασφάλεια δικαίου τέλο πάντων, ε, η απαγόρευση της αυθαιρεσίας, κακοδικίας, τα της εκτελεστικής εξουσίας, η αντικειμενικών δικαστηρίων, οπότε όλα αυτά αφορούν και το ότι οι γυναίκες έχουν φυγεί όσον αφορά βασικά δικαιώματα στην υγεία και στην αναπαραγωγή και έχουμε και επιδείνωση κατάσταση για τις μη οργανώσεις και όπως είπαμε θα μπορέσουν αν θέλουν οι αρχές της χώρας να συμμετάσχουν στην παρουσίαση της έκθεσης αρχάς του Δεκεμβρίου. Και ξεκινούμε τώρα την ακρόαση. Πρώτο πάνελ θεσμικά όργανα, πρόσωποι των θεσμικών οργάνων, ο πρώτος αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Φρανς Τίμερμαντς. Έχει στη διάθεσή του 15 λεπτά. Φρανς, um, Ευχαριστώ πάρα πολύ και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας που οργάνωσε την σημερινή ακρόαση για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Πολωνία και ειδικά όσον αφορά την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Σας ευχαριστώ για την πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση που μας δώσατε για την επίσκεψή σας στην Πολωνία που νομίζω ότι ευθυγραμμίζεται και με τις ανησυχίες που είχα εκφράσει εξ ονόματος Κομισιόν ήδη πολλές φορές. Αν μου επιτρέψετε τώρα θα σας ενημερώσω για το που βρισκόμαστε και ποιες είναι οι βασικές εξελίξεις από την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε στις 28 Ιουνίου. Να επενθυμίσω τις βασικές ανησυχίες ε, της ε, Κομισιόν. Αφορούν τις μεταρρυθμίσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου, του Εθνικού Συμβουλίου Δικαιοσύνης, ε, τους τακτικούς δικαστές, το πειθαρχικό καθεστώς, ε, τους ε, πρόεδρους των δικαστηρίων ε, και την σύνθεσή τους. Η κυρία σκέψη της Κομισιόν όταν ενεργοποιήσαμε το άρθρο 7 τον Δεκέμβριο του 2017 ήταν το σορευτικό και συστημικό αποτέλεσμα των διάφορων αυτών μεταρρυθμίσεων στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνη και την διάκριση των εξουσιών το κοινό μοτίβο που υπάρχει είναι ότι η νομοθετική και η εκτελεστική εξουσία μπορούν τώρα να εμπλακούν σε ολόκληρο το φάσμα της δικαιοσύνης. Και λυπούμε ε, για το ότι μέχρι σήμερα καμία από τις σχετικές ανησυχίες στην αιτιολογημένη πρόταση της Κομισιόν δεν έχει απαντηθεί από τις πολωνικές αρχές και εξακολουθεί να υπάρχει συστημικός κίνδυνος για το κράτος δικαίου. Τώρα θα ήθελα επίσης να αναφέρω κάποιες νέες ανησυχητικές εξελίξεις. Εν τω μεταξύ, η πειθαρχική λειτουργή του Υπουργείου Δικαιοσύνης έχουν ξεκινήσει μια σειρά προκαταρκτικών πειθαρχικών έρευνων καταδικαστών που συμμετείχαν σε δημόσιες συζητήσεις, έκαναν δημόσιες δηλώσεις για τις μεταρρυθμίσεις ή είχαν παραπέμψει κάποια αιτήματα στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, σε κάποιες περιπτώσεις η πειθαρχική αυτή λειτουργεί ρητός αρνήθηκαν ότι οι δικαστές ε, αρνήθηκαν οι δικαστές τους οποίους ερευνούσαν να έχουν μαζί τους τους νομικούς τους συμβούλους. Παραπέμπω εδώ πέρα στην ανακοίνωση της ε, πέντε ενώσεων πολωνών δικαστών που αναφέρονται συγκεκριμένα σε εκφοβισμό των δικαστών που ζήτησαν μια προκατακτική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Και είχαμε ε, βεβαίως ε, τέτοια αιτήματα από τα πολωνικά δικαστήρια. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πέντε τέτοια προδικαστικά ερωτήματα που έχουν αποσταλεί από το ανώτο δικαστήριο και τρία προδικαστικά ερωτήματα από τα τακτικά δικαστήρια. Τα περισσότερα από αυτά τα ερωτήματα αφορούν ακριβώς τις ανησυχίες της ε, Κομισιόν που υπάρχουν στην αιτιολογημένη πρότασή μας. μια πρώτη περίπτωση το δικαστήριο αποφάσισε να δεχτεί το αίτημα για μια ταχεία εκδίκαση και όρισε την ακρόαση στις 12 Φεβρουαρίου του 2019. Αυτό το οποίο είναι ακόμη πιο ανισχυτικό είναι ότι ως αντίδραση σε αυτές τις παραπομπές έγιναν διάφορες δηλώσεις από την εκτελεστική εξουσία και ζητήθηκε μάλιστα από ένα δικαστήριο να αποσύρει το προδικαστικό το ερώτημα. Όσον αφορά την κατάσταση του Πολωνικού Ανωτάτου Δικαστηρίου, έχει υπάρξει μια επιτάχυνση της εφαρμογής ε, του καθεστώτος συνταξιοδότησης, παρά το ότι αποφάσισε στις 2 Αυγούστου το δικαστήριο να ανασταλούν οι σχετικές διατάξεις και να παραπεμφθεί το ζήτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αγνόησε την σχετική απόφαση και απέρριψε το αίτημα παράτασης ε, που υπέβαλαν 7 δικαστές που επηρεάζονταν από την χαμηλότερη ηλικία συνταξιοδότησης και 15 δικαστές ήδη ε, θεωρούνται συνταξιοδοτηθέντες. Ως αποτέλεσμα αυτού, 22 από τις 27 δίκαστες του ανωτάτου δικαστηρίου που επηρεάζονται από το νέο όριο ηλικία θεωρούνται ως συνταξιοδοτηθέντες. Αυτό περιλαμβάνει και τον πρώτο πρόεδρο του ανωτάτου δικαστηρίου, η θητεία του οποίου προστατεύεται συνταγματικά και κανονικά πρέπει να λήξει το 2020. Όπως ξέρετε, στις 24 Σεπτεμβρίου η Κομισιόν αποφάσισε να παραπέμψει την Πολωνία στο ΔΕΚ ε, ε, με μια διαδικασία επί παραβάση για το καθεστώς συνταξιοδότησης των δικαστικών. Κατόπιν αυτού του αιτήματος, ο αντιπρόεδρος του δικαστηρίου στις 19 Οκτωβρίου αποφάσισε να διατάξει προσωρινά μέτρα για να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία του ανατάτου δικαστηρίου. Τα προσωρινά μέτρα που διέταξε το δικαστήριο και άρχισαν να ισχύουν αμέσως προσωρινά ικανοποίησαν όλα τα αιτήματα της Κομισιόν. Την Παρασκευή που μας πέρασε υπήρξε μια ακρόαση ενώπιον του δικαστηρίου και επί τη βάση της οποίας θα ληφθεί η τελική απόφαση επί των αιτημάτων της Κομισιόν. Χτες, σύμφωνα με την προσωρινή διαταγή, η Πολωνία έδωσε στην ε, Κομισιόν μια έκθεση όσον αφορά το καστός της εφαρμογής και αυτή τη στιγμή αναλύουμε την έκθεση αυτή. Μετά από την έντολη ε, του δικαστηρίου, ο πρώτος πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου συγκέντρωσε όλους τους δικαστές που επηρεάζονται από τον όριο ηλικία για να παρουσιαστούν στα καθήκοντά τους. Και οι 22 εμφανίστηκαν και ήδη του έχουν ανατεθεί υποθέσεις. Είναι μάλιστα σημαντικό οι δικαστές αυτοί να συνεχίσουν να δικάζουν με πλήρη ανεξαρτησία εν αναμονή των περαιτέρω αποφάσεων του Δικαστηρίου της Ένωσης. Σημειώνουμε λοιπόν με ανησυχία το ότι η πολωνική κυβέρνηση θεωρεί ότι απαιτείται μια νομοθετική αλλαγή για τη συμμόρφωση με την απόφαση του δικαστηρίου για να επιστρέψουν οι δικαστέ στα καθήκοντά του. Ε, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει προτείνει κάτι τέτοιο μέχρι σήμερα. Επίση, σημειώνω με ανησυχία ένα πρόσφατο ψήφισμα του νέου Εθνικού Συμβουλίου για την Δικαιοσύνη που λέει ότι εν λόγω δικαστές είναι ακόμα σε καθεστώ συνταξιοδότηση. Οπότε τίθεται ένα αμφιβόλο ικανότητα του Εθνικού Συμβουλίου να διασφαλίσει την εξαρτησία τη δικαιοσύνη. Να υπενθυμίσω ότι στι 17 Σεπτεμβρίου το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δικαστικών Συμβουλίων είχε αποφασίσει να αναστείλει την ε, συμμετοχή της σχετικής πολωνικής αρχής. Αυτά τα μέτρα πρέπει να τα δούμε σε ένα γενικότερο πλαίσιο που περιλαμβάνει και το συνταγματικό δικαστήριο τον Οκτώβριο. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης ε, ζήτησε να κηρυχθεί παράνομη παράνομος ο σχετικός μηχανισμός στην περίπτωση που αφορούσε ακριβώς την μορφή και οργάνωση του πολωνικού συστήματος δικαιοσύνη. Το αίτημα αυτό αντιβαίνει ε, στις ε, θεμελιώδεις αξίες της Ένωσής μας. Ολόκληρο το σύστημα δικαιοσύνης Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίζεται σε πλήρη και ανεμπόδιστη πρόσβαση στο ΔΕΚ από τα εθνικά δικαστήρια. Δεν θα πρέπει να παρεμβαίνουν άλλες αρχές σε αυτήν την πρόσβαση. Όσον αφορά λοιπόν το συνταγματικό δικαστήριο, προσφάτως ο Πολωνός συνήγορος του πολίτη είπε πως η σύνθεση του δικαστηρίου σε μια πολιτικά ευαίσθητη υπόθεση άλλαξε πάλι χωρίς επαρκή αιτιολόγηση και προσθέθηκε ένας επιπλέον δικαστής. Και έτσι απέσυρε την υπόθεση ο διαμεσολαβητής. Δυστυχώ. δεν μπορώ να σε ενημερώσω σήμερα για κάποιες θετικές εξελίξεις. Έτσι είναι σοβαρή η ανάγκη να αλλάξει πορεία η πολωνική κυβέρνηση και να ανταποκριθεί πλήρως σε όλες αυτές τις ανησυχίες. Το δικαστήριο θα λάβει μια οριστική απόφαση κάποια στιγμή το 2019 για τις υποθέσεις οι οποίες βεβαίως δεν έχουν παραπέμφθει στο 10 η Κομισιόν παραμένει στην διάθεση της ε, Πολωνίας για να λυθούν αυτά τα ζητήματα με διάλογο. Να το ξαναπώ. Η Κομισιόν θέλει διάλογο με την πολωνική κυβέρνηση για να επιληθούν αυτά τα ζητήματα. Αυτό είναι ο ευρωπαϊκός τρόπος με διάλογο. Αλλά η Κομισιόν είναι επίσης θεματοφύλακα των συνθήκων πρέπει να φροντίσουμε η διάκριση των εξουσιών να είναι εγγυημένη. Είναι βασική αρχή της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όπως και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Κομισιόν αναγνωρίζει το δικαίωμα του κάθε κράτους μέλους να μεταρρυθμίσει την δικαιοσύνη, αλλά η μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης δεν μπορεί να οδηγεί στο να καταργηθεί η διάκριση των εξουσιών και να υπάρχει μια δικαιοσύνη υπό πολιτικό έλεγχο. Δεν μπορεί να είναι αυτό το αποτέλεσμα. Αλλά δεν αμφισβητούμε το δικαίωμα των πολωνικών αρχών να κάνουν μεταρρυθμίσει. Και πάλι θα το ξαναπώ. Θέλουμε να επιληθεί αυτό το ζήτημα με διάλογο, με βάση την ε, αιτιολογημένη ε, άποψή μας. Λοιπόν, καταλήγοντας, θα ήθελα να πω πώς η υπεράσπιση του κράτου δικαίου είναι κοινή ευθύνη όλων των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και είναι σημαντικό η Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά και να προσθέσω και το Συμβουλίο ο οποίο στην διαδικασία του άρθρου 7 έχει μία ιδιαίτερη ευθύνη. Οπότε, θα ήθελα ακόμη μια φορά να επαναλάβω την έκκλησή μου στην πολωνική κυβέρνηση να μας βοηθήσει να λύσουμε αυτό το ζήτημα ε, επί τη βάση των αρχών που αναφέρονται στην συνθήκη στο άρθρο 2. Αυτοί είμαστε ως Ευρωπαίοι. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να προχωρήσουμε σε αυτό το ζήτημα. Σεβόμενοι το κράτος δικαίου, την διάκριση των εξουσιών και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Αυτό είναι δικαίωμα του κάθε Πολωνού πολίτη. Γιατί ε, μην ξεχνάμε αυτό το οποίο είπε και ο πρόεδρός σας. Ε, όταν ε, δικάζει με βάση το κοινοτικό δίκαιο, ένας πολωνός δικαστής είναι και ευρωπαίος δικαστής και αντιστρόφως όταν κρίνει αυτά τα ζητήματα ένας δικαστής ε, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι και πολωνός δικαστής. Είναι λοιπόν ενιαίο το νομικό μας σύστημα και θα πρέπει να διατηρήσουμε την διάκριση των εξουσιών για να λειτουργήσει η ένωμη Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Επίτροπε. Τώρα. Κανονικά θα μεσολαβούσε η κυβέρνηση να εξηγήσει. δυστυχώ η πολιτική κυβέρνηση δεν απέστειλε εκπρόσωπο για τους λόγους που εξήγησα. Οπότε, προχωρούμε στην πρώτη συνεδρία ερωτήσεων απαντήσεων μετά την ομιλία του Επιτρόπου. Κάποια από τα μέλη της υποστολής στην Βαρσοβία θα λάβουν τον λόγο. Να πω ότι κάποιοι αποσιάζουν για διάφορους λόγους από την Επιτροπή που επισκέφθηκε την Πολωνία. Ο κύριος Τομασεύσκη, όχι, Άγγελ, Κύριο Σέγγελ, παρακαλώ. Πρώτος, από το ΕΛΚ. Μέλος της αντιπροσωπείας από το ΕΛΚ. Κλώδη, ευχαριστώ. Θα είμαι μάλλον σύντομος. Διότι οι περιστάσεις δυστυχώς επιβεβαιώνουν αυτά που πιστεύουμε εδώ και μήνες. Η υποστολή... Στην Πολωνία έλαβε χώρα σε εποχή που η κυβέρνηση και οι αρχές πίστευαν ότι το παρακάνουμε. Ε, δεν είχαμε πάει να διαπιστώσουμε κάτι παραπάνω από την απλή πραγματικότητα. Το σίγουρο είναι ότι δεν γίναμε δεκτοί πολύ φιλικά. Συζητούμε λοιπόν σήμερα ένα θέμα χωρί τις πολιτικές αρχές. Ούτω ή άλλω δεν ήταν διαρρυθμένοι να κάνουν κάποιε προχωρήσει να μιλήσουν, να συζητήσουν και δυστυχώς αυτό επιβεβαιώνεται και σήμερα. Δεν νομίζω ότι μπορούν να χειροτερέψουν περισσότερο τα πράγματα. Το βέβαιο είναι ότι οι πολωνικές αρχές δεν έχουν καμιά όρεξη για διάλογο με την Κομισιόν, ούτε πριν υπήρχε, ούτε υπήρχε τέτοια βούληση τον Σεπτέμβριο όταν επισκεφθήκαμε την Πολωνία. Και δεν εκπλησόμεθα και με τη σημερινή στάση των πολωνικών αρχών. Σε κάθε περίπτωση, οφείλουμε να συνεχίσουμε να προσπαθούμε να πείσουμε τις πολωνικές αρχές ότι αυτό είναι λάθος θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να πείσουμε και την κοινή γνώμη στην Πολωνία ότι νοιαζόμαστε για την Πολωνία και ότι συνεχίζουμε να προσπαθούμε. Δεν θα καταλήψουμε την προσπάθεια. Θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε σε όλα τα μέτωπα. Στις τελευταίες εκλογές στην Πολωνία είχαμε ενδεχομένω μία μικρή ένδειξη ότι τα πράγματα μπορεί να αλλάζουν. Δηλαδή, ενδέχεται κάποιοι εντάξει, του πολωνικού λαού να αντιλαμβάνονται ότι η πολωνική κυβέρνηση βαδίζει σε δρόμο που δεν είναι ο σωστός. Κάποιοι λοιπόν μάλλον το αντιλαμβάνονται. Η Πολωνία πρέπει να μείνει μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας, προσκολλημένη στις αξίες και τις πεπιθήσεις που συμμεριζόμαστε. Και σίγουρα στις αρχές αυτές δεν ανήκει η υποδούλωση της δικαιοσύνης. Και πρέπει, όπως είπατε ο Κλοντ και ο Επίτροπος, πρέπει να συνειδητοποιήσει και η Πολωνία ότι το σωρευτικό αποτέλεσμα των μέτρων που έλεγε η πολωνική κυβέρνηση είναι μια πλήρω πολιτικοποιημένη δικαιοσύνη. Περί αυτού πρόκειται. Πολιτικο, πλήρω πολιτικοποιημένη δικαιοσύνη. Και αυτό είναι απαράδεκτο. Ευχαριστώ. Και τώρα, άλλο ένα μέλο τη αντιπροσωπεία. Σπινέλη, και Σπινέλη από την Παρακαλώ. Μπάρμπρα, έχει τον λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον Αντιπρόεδρο Τίμερμανς για τα όσα μας παρουσίασε. Ήμουν στην Πολωνία στη διάρκεια της αποστολής μας. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό για τους δικαστές με τους οποίους ε, συναντηθήκαμε για το τι θα κάνει ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Κοινοβούλιο. Πραγματικά υπάρχει ε, αγωνία, υπάρχουν προσδοκίες για το μήνυμά μας ή της Κομισιόν. Τώρα όσον αφορά το άρθρο 7. Δεν ξέρω αν συμφωνούν και έχουν την ίδια εντύπωση με εμένα οι συνέλφοι που ήταν μαζί εκεί, αλλά περισσότερα περιμένω από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο παρά από το άρθρο 7 και όχι γιατί το 7 δεν το θεωρούν σημαντικό. θεωρείται κάτι πολύ θετικό το ψήφισμά μας σχετικά, αλλά από πλευράς αποτελεσματικότητας και από πλευράς δυνατότητας του να περάσει το μήνυμα και για αυτούς είναι φάρος ελπίδας το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Κύριε την Πρόεδρε, θα ήθελα να σας πω το εξής. Καταλαβαίνω απολύτω ότι εσείς έπρεπε να περιοριστείτε στα νομικά γιατί αυτές είναι οι αρμοδιότητές σας και επίσης σχολιάσατε το δικό μας ψήφισμα. Όμως, κράτος δικαίου είναι ένα όραμα, μία αρχή που περιέχει και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Οπότε πάντα σε σχέση με την αποστολή μας στη χώρα, τι είδα. Και ο πρόεδρος, ο πρόεδρος μας που προείδευε της αποστολής Μωράς θα το παρατήρησε ότι πολλά είναι τα δικαιώματα τα οποία κινδυνεύουν. Η ελευθερία του τύπου και άλλα και αναφέρομαι και στα αναπαραγωγικά δικαιώματα. Γιατί έχουμε εκείνο το νομοσχέδιο το σχετικό το οποίο ευτυχώς δεν πέρασε στην ακραία του μορφή όπως ήθελε η κυβέρνηση. Όλα αυτά η απειλή ακόμα υπάρχει. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος της Εκκλησίας. Το οποίο φυσικά δεν ε, προβλέπεται από το Σύνταγμα. Όμως εμείς ακούσαμε σχετικά όλους τους ε, φορείς που ασχολούνται με τα πολιτικά δικαιώματα. Um, Ευχαριστώ κύριε Σπινέλη. Και τώρα οι συνάδελφοι με τη σειρά που έχουν δηλώσει την πρόθεση τους να μιλήσουν ως πρόεδρος της αποστολής να πω κάτι για αυτό το οποίο είπε ο κύριος Άγγελ σχετικά με τη θέση δηλαδή, του Κοινοβουλίου στην Βαρσοβία. Τονίσαμε, νομίζω και θα το επιβεβαιώσουν δύο από τα μέλη που είναι εδώ σήμερα μαζί μας, ότι δεν είναι πρόκειτο για διεπιστορική των πραγμάτων επιτροπή, Αυτό το καταστέμε σαφές προς τις πολωνικές αρχές, προς όλους τους συνομιλητές μας, που ήταν εκεί για το συγκεκριμένο σκοπό. Πρέπει να καταλάβουν και οι συναδελφοί ποιος ήταν ο ρόλος μας σε αυτόν τον μηχανισμό, ένα πολύ συγκεκριμένο μηχανισμό. Είναι στο πλαίσιο του διαλόγου, όπως είπε και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, ο κ. Επίτροπος. Και εμεί θέλουμε να έχουμε ένα διαρκή διάλογο με την Πολωνία και τις πολωνικές αρχές, επί θεμάτων κράτους δικαίου. Υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία λοιπόν. Μπόνι, παρακαλώ. Θα μιλήσω πολωνικά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το κλιμάκιο που μετέβη στην Πολωνία. Ευχαριστώ για το έργο σας. Περιμένω την έκθεση βεβαίως για να μπορέσω να συνεχάγω μερικά συμπεράσματα. Ευχαριστώ και τον Τύρο Τίμερμανς για την συνεπή παρουσίαση των θέσεών του και την ερμηνεία των γεγονότων. Αυτό που έκανε η Κομισιόν ήταν πολύ σημαντικό. Ζήτησε από τον Υπουργό Δικαιοσύνη, να λάβει μέτρα, γιατί το θέμα είναι και νομικό και πολιτικό. Για όσου πιστεύουν σήμερα ότι όλα αυτά αποσκοπούν στην επίκριση της Πολωνίας και γιατί είναι δυνατόν όλοι να είμαστε μαζί. Τι, τι να σου πω, τα πράγματα είναι πολύ απλά. Το πρώτο πράγμα είναι ότι υπάρχει μια εντολή του δικαστηρίου, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου προς την πολωνική δικαιοσύνη. Δεύτερον, εμείς συνεργαζόμαστε με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Αντιθέτως, η έλλειψη συνεργασίας είναι αυτό το οποίο χαρακτηρίζει το Πολωνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης. Και δείτε, ε, στην Ουγγαρία συμβαίνουν αντίστοιχα, αλλά οι Ούγγροι ήρθαν εδώ, το Ουγγρικό Υπουργείο Δικαιοσύνης ήρθε να μιλήσει. Εν συνεχεία έχουμε συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά το κράτος δικαίου, τις οποίες προωθούμε. Θα ήταν αδιανόητο μετά να αμφισβητήσουμε αποφάσεις του συνταγματικού δικαστηρίου. Κάθε πολιτισμένη χώρα έχει συνταγματικό δικαστήριο. Λοιπόν, δεν μπορεί κανείς να κατεδαφίζει τους θεσμούς και δι της δικαιοσύνης σε καμία χώρα. Δεν μπορεί κανείς λοιπόν να πολιτικοποιεί τη δικαιοσύνη. Αυτά είναι μάλλον σημάδια της προσπάθειας να κατακτήσει κανείς την εξουσία από όλες τις πλευρές. Γιατί δεν είναι μόνο δικαιοσύνη, είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι η κοινωνία των πολιτών. Κάποιοι θέλουν να τα καταλάβουν όλα. Κάποιοι θέλουν να ελέγξουν ακόμα και την ελεύθερη αγορά. Κάποιοι θέλουν να ελέγξουν τις χρηματοπιστωτικέ αγορές. Συνεπώ ναι, ήρθε η ώρα να κάνουμε κάτι. Α αξιοποιήσουμε αυτήν την απλή συνταγή, θα έλεγα, Ζητώντα πολύ απλά να σταματήσουν οι παραβάσεις του ευρωπαϊκού, του κοινοτικού δικαίου. Μπορεί να διαφωνεί κανεί ε, σε πολλά με την Ευρώπη, αλλά εδώ δεν νομίζω ότι χωράει αφιβολία. Βιόρκ παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που ήρθατε μαζί με τους ε, συναδέλφους μου μια ομάδα που λεγόμαστε Όλοφας σας απευθύνα μια επιστολή, δεν απαντήσατε θέλω όμως να την επαναλάβω γιατί όταν μιλάμε για το κράτος δικαίου πρέπει να δούμε το ποιος είναι ο στόχος και το θύμα όταν δεν υπάρχει κράτος δικαίου θα αναφέρω δύο παραδείγματα που αναφέραμε στην επιστολή μας παραδείγματος χάρη στο συνταγματικό δικαστήριο εξετάζουν τώρα το εάν είναι συνταγματική η έκτρωση, η οποία επιτρέπεται μόνο όταν υπάρχει σοβαρή ζημιά στο έμβριο. Έτσι είναι το 90% των εκτρώσεων. Το άλλο είναι μια περίπτωση διάκρισης ε, ΛΟΑΤΚΙ που ε, κρίθηκε στα κατώτερα δικαστήρια υπέρ της ε, σχετικής ε, κοινότητας. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος είναι και Γενικός Αγγελέας, θα ασκήσει έφεση στο συνταγματικό δικαστήριο. Λοιπόν, όταν μιλάμε για το κράτος δικαίου στην Πολωνία πρέπει να δούμε τις συγκεκριμένες συνέπειες στη ζωή των ανθρώπων. Οπότε, όταν μιλάμε εδώ για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμείς ε, τα έχουμε τονίσει όλα αυτά στην έκθεσή μας και θα πρέπει και εσείς ακριβώς να τα παρακολουθείτε και ε, να γνωρίζετε ποιους στοχεύει αυτή η έλλειψη ανεξαρτησία δικαιοσύνη. Γιατί υπάρχει και η Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και το άρθρο 2 τη συνθήκη. Σα ευχαριστώ, κύριο Γιούρεκ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, ήλπιζα ότι θα πάρει λόγο αμέσως μετά τα μέλη της ε, αντιπροσωπείας, αλλά αποκλείστηκα γιατί από φαίνεται ένας Πολωνός βουλευτής ε, δεν μπορεί να συζητήσει με τις πολωνικές αρχές. Ευτυχώς βεβαίως δεν στάθηκε αυτό ικανό να με σταματήσει. Τα συζήτησα αυτά με τον Πολωνό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορείτε να ε, τα συζητήσετε κι εσείς ε, μαζί του. Λοιπόν, να σας πω τώρα, να περάσω τώρα στην ουσία. Υπάρχουν κάποιες επικίνδυνες εξελίξεις όσον αφορά την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και των πολωνικών δικαιωμάτων στην συζήτηση αυτή. Ελπίζω να ακούσω την ε, δική σας ε, την θέση, την θέση του κύριου Τίμερμανς. Όπως γνωρίζει ο κύριος Τίμερμανς και οι περισσότεροι εξημών τι μας ενδιαφέρει, η συζήτηση αυτή έχει ήδη οδηγήσει σε κάποιες ε, περιπτώσεις όπου δεν εκτελέστηκαν κάποια εντάλματα σύλληψης με βάση κάποιες αυθαίρετες αποφάσεις ε, κρατών μελών. Παραδείγματος χάρη από την Ιταλία. Ένας Ιταλός δικαστής ε, αρνήθηκε να κάνει κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε, ε, το θέμα της πολιτικής ελευθερίας δεν αφορά μόνο τη σχέση μεταξύ κρατών. Η ελευθερία είναι πρώτα απ' όλα και το να να φροντίζουμε τους ε, πολίτες μας. Ε, και οι οι πολίτες έχουν δικαίωμα να διώκονται οι εγκληματίες και να αισθάνονται ασφαλείς. Όλοι γνωρίζουμε ότι και τα κράτη-μέλη, όχι μόνο η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο, μπορούν, ε, σύμφωνα με την συνθήκη, να κατηγορούν αλλήλους σε σχέση με την ε, ορθή λειτουργία του άρθρου 2. Το γεγονός ότι 10 κράτη-μέλη κατηγορούν 10 άλλα κράτη-μέλη σημαίνει ότι ε, μπορούν να μην πληρούν τις συμβατικές τους ε, υποχρεώσεις. Νομίζω ότι θα ήταν ένα δείγμα αμεροληψίας εάν ο πρόεδρος της Κομισιόν, εξαρτήτως της προσωπικής του γνώμης, αντιδρούσε. Γιατί βεβαίως το πρώτο καθήκον του ε, πολωνικού κράτους είναι να προστατεύει τους πολωνούς πολιτές από τους εγκληματίες. Η συζήτηση λοιπόν αυτή δεν αφορά μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Κομισιόν και τις πολωνικές αρχές, αλλά είναι μια επίθεση κατά της ε, πολωνικής ε, κοινωνίας και του πολωνικού δικαίου. Εγώ σέβομαι την συνάδελφο, την Μπάρμπαρα Σπινέλη, αλλά ε, μου προξένει σε έκπληξη αυτό το οποίο μόλις είπε. Ο νόμος αυτός είναι ακόμα σε ένα επίπεδο πρωτοβουλίας ε, που στόχο έχει να σταματήσει τις εκτρώσεις και όμως υπάρχει ήδη ένας αντίκτυπος ε, στα δικαιώματα της ε, Πολωνίας. Το κίνημα αυτό ήταν μια πρωτοβουλία των πολιτών. Και ο πρόεδρος, ο Κλοντ Μωραές, εξέφρασε τη λύπη του για το ότι δεν υπάρχουν εκπρόσωποι των πολωνικών αρχών. Και εγώ λυπάμαι για το ότι δεν υπάρχουν εκπρόσωποι της εν λόγω πρωτοβουλίας. Ζήτησα να έρθει εδώ πέρα η κυρία Καγιακόντεκ, η οποία ε, είναι η νόμιμη εκπρόσωπος και ζήτησε να έρθει εδώ και πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί δεν ήρθε δεν σεβόμαστε εδώ πέρα το δικαίωμα του συνεταιρίζεστε και ακριβώ ε, και την κοινωνία των πολιτών. Και λυπούμε γι' αυτό. Και πραγματικά δεν μου άρεσαν αυτά τα οποία είπε η κυρία Σπινέλη για την ε, Εκκλησία, η οποία αποτελεί μέρος της κοινωνίας ε, των πολιτών, όπως και τα ΜΜΕ και η επιστημονική κοινότητα. Έτσι γίνεται πιο πλούσια η κοινωνία, όλοι έχουμε δικαίωμα να λάβουμε μέρος στην συζήτηση αυτή και να εκθέσουμε τα επιχείρηματα μας. Δεύτερον, όταν μιλάει για το πολωνικό δίκαιο, κυρία Σπινέλη. κοιτάξτε, να σας πω ότι το προήμιο του συντάγματο ε, λέει ότι είμαστε γνώμονες κτλ. Αλλά επίση λέει ότι θα πρέπει να ε, γίνει και διάλογο ε, με τι θρησκευτικέ αρχέ και δεν ξέρω το, τι, το εάν το κάνει αυτό όντως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι περίεργο να ασκούμε κριτική επειδή λέει η πολωνική κοινωνία κάνει κάτι τέτοιο. Ε, σκέφτομαι και αυτό το μόνιμο πραξικόπημα που έλεγε ο Μίτεραν. Υπήρχαν ε, συνεχείς αναταραχές ε, και ο Φρανσό Μιτεράν είχε πει πως κάποιοι δεν οροδούν προδενός για να πετύχουν τον στόχο τους και ανέφερε τον, τα λόγια του Μισελ Ντεμπρέ μίλησε εκείνος για τον νομικισμό ο οποίος δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες ε, του κράτους. Όταν έγινε αυτό, όταν ο Ντεγκόλ υπέγραφε τις ε, συνθήκες των ηλισίων. Ε, λοιπόν, αυτές οι συγκρίσεις δεν είναι επιχειρήματα. Απλά θέλω να πω ότι δεν πρέπει να υπάρχουν αυτές τις διχοτομίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συζήτηση όλων αυτών των πραγμάτων επίσης υπάρχουν και στην Πολωνία και δεν μιλάμε για εξωτερικές ε, πιέσεις. Και το τελευταίο μου σχόλιο προς τον πρόεδρο. Η Κομισιόν είναι θεματοφύλακα των συνθήκων και η συνθήκη λέει ότι θα πρέπει να φροντίζουν για την εφαρμογή τους. Αλλά θα πρέπει να υπάρχει και διάκριση των εξουσιών. Ας περιμένουμε λοιπόν την απόφαση του δικαστηρίου. Η Κομισιόν λοιπόν δεν είναι κάποια η οποία μπορεί να διατάξει κάποιον και αν δεν υπάρχουν επιχειρήματα δεν πρέπει να λάβουν υπόψη τις ε, θέσεις της. Η κυρία Μπαρβαρα Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν έλαβα μέρος στην αποστολή στην ε, Πολωνία. Έτσι είχαμε συμφωνήσει. Να μην πάμε η Πολωνία στην Βαρσοβία. Η σκοπό με αντικειμενικό τρόπο να προσπαθήσει να μαζέψει κάποια στοιχεία εκεί. Πάντως υπάρχει κάτι που με προβληματίζει. Τώρα που άκουσα και τον κύριο Γιούρεκ μας μίλησε για τις μεταρρυθμίσεις του Ντεγκόλ. Μα γιατί να έχουμε πολιτικές αλλαγές. Γιατί να έχουμε μεταρρυθμίσεις στη δικαιοσύνη και αλλού. Οι αλλαγέ στην Πολωνία έγιναν για να είναι πιο αποτελεσματικές διαδικασίες. Όχι. Τώρα οι διαδικασίες είναι, κρατάνε περισσότερο. Είναι πιο επαγγελματική τώρα η διαχείριση των πραγμάτων. Όχι. Ένα σώρο άτομα χωρίς ικανότητες τώρα δικάζουν Όλα αυτά έγιναν για να είναι πιο δίκαιες οι δίκες. Όχι, γιατί τώρα έχουμε περισσότερα ενδικά μέσα κατά των αποφάσεων. Των αποφάσεων σε πρώτο βαθμό. Άρα για κάποιο άλλο λόγο είναι αυτές οι αλλαγές και δεν είναι τόσο δύσκολο κανείς να καταλάβει ποιος ήταν ο σκοπός. Όλα αυτά έγιναν για να αλλάξουν τα πρόσωπα που υπηρετούν τη δικαιοσύνη. Το πειθαρχικά... Οι αλλαγέ στο πειθαρχικό τμήμα του Ανατότου Δικαστηρίου ήθελαν να βάλουν τους δικούς τους παντού. Ήθελαν να ελέγξουν και τους δικαστές που δεν αντικαταστάθηκαν. θέλουν να τρομάξουν αυτούς που παρέμειναν με τα πειθαρχικά. Και τα ακούσαμε αυτά σήμερα και από τον κύριο Τίμερμαντς. Ότι υπάρχουν πειθαρχικές διαδικασίες κατά δικαστών. Οι δικαστές αυτοί δεν δικαιούνται συνηγόρου σε αυτές τις πειθαρχικές διαδικασίες. Και έτσι η Ευρώπη γίνεται μάρτυρας σκανδάλων διαφθοράς στη χώρα. Αυτά σχετικά με την εποπτεία της εθνικής οικονομίας. Και ένα στιγμή της τράπεζας κατηγορείται για δωροδοκία. Οπότε γι' αυτό και υπήρχε η πρόθεση ελέγχου της δικαιοσύνης. Πάει η διέρεση των εξουσιών. Όλοι να ελέγχονται στενά. Έτσι, κάποιοι που διαπράττουν εγκλήματα να είναι στο απειρόβλητο. και η στάση της χώρας, της κυβέρνησης, έναντι του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, δείχνει το ότι η κυβέρνηση δεν είναι καλόπιστη. Ο πρόεδρος. Στις 3.30 πρέπει να φύγει ο πρόεδρος. Άρα μην με Κάποιος μίλησε επί 8 λεπτά. Όλο και περισσότεροι ζουν το λόγο, οπότε παρακαλώ συνάδελφοι, περιοριστείτε σε ένα δίλεπτο. Ο επόμενος. Ο κύριος Dialog bereit ist. Da müsste man aber zunächst einmal diskutieren, was für ein ναι, συμφωνώ, αλλά θα έπρεπε να συζητήσουμε πρώτα απ' όλα το τι είδου ε, διάλογος είναι αυτός. Είναι ένας διάλογος με ανοιχτό αποτέλεσμα. Όχι. Απλά αναμένουμε από τους ε, προσκεκλημένους ε, να συμμορφωθούν με κάποια πράγματα και όταν μιλάμε για ανεξαρτησία των δικαστών έχω όλο και περισσότερο την εντύπωση ότι εννοείται ακριβώς ε, την υποταγή των δικαστών στις αμφίβολες αυτές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που είναι και τεχνητές ε, αξίες και έχουμε μια χριστιανική χώρα όπως η Πολωνία όπου δεν είναι αυτονόητο να συμφωνήσουν με τη δολοφονία ενός παιδιού με στο σώμα της ε, μητέρας του ή να συμφωνήσουν με τον γάμο των ομοφιλοφιλών. Αυτό απλά πρέπει να το δεχτείτε. Σε άλλες χώρες ο κόσμος έχει άλλες αξίες. Και εδώ μέσα βεβαίως πάντα γίνεται ο αγώνας ε, να υπάρξει παραχώρηση όλων αυτών ε, των αξιών που πιστεύουν οι μουσουλμάνοι, αλλά αρνείστε το ίδιο στου ε, χριστιανού. Οι χριστιανοί όμω δημιούργησαν την Δύση και μας έκαναν αυτό το οποίο είμαστε σήμερα. Εάν ε, ασκείται κριτική στην ανεξαρτησία τη δικαιοσύνη, γιατί έπεσε το όριο συνταξιοδότηση από τα 70 στα 65, αυτό δείχνει το πόσο πολύ παρεμβαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα κυρίαρχα δικαιώματα ενό κράτου. Και ελπίζω μόνο η Πολωνία να συνεχίσει τις ε, προσπάθειες της ε, και να αποτύχουν ε, όλα αυτά τα σχέδια του Σόρους. Γιατί κάπου θα πρέπει να έχει δικαίωμα να συνεχίσει και να υπάρχει η χριστιανική δύση στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Επιτρόπος είπε ότι θα ήθελε να φύγει στις 3.30. Λοιπόν, να ακούσουμε τώρα τις κυρία Σόφη Ινετφέλτ και την κυρία Βυσνιεύσκα. Η κυρία Σόφη Νετφέλτ. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πέρα από το περιεχόμενο της παρέμβασης ε, του κύριου Γιούρεκ, ε, δεν είναι νομίζω τρόπος αυτός αντιμετώπιση των συναδέλφων να μιλάτε τόσο πολύ και να μην αφήνετε χρόνο για τους υπόλοιπους αλλά για το θέμα αυτό, το είπε και ο κύριος Βόιτ ε, μόλις τώρα, γιατί εδώ πέρα έχουμε μια τελείως διαφορετική ατζέντα. Δεν είναι τεχνικό το ζήτημα ε, για τις ε, μεταρρυθμίσεις ακριβώς, είναι κάτι το τελείως διαφορετικό. Να καταστραφούν τα δικαιώματα των γυναικών, των ΛΟΑΤΚΙ, του πλωραλισμού, της ελευθερίας, της και τελικά της ε, δημοκρατίας. Η ατζέντα αυτή έχει όνομα. Υπάρχει ένα μανιφέστο με τίτλο «Αποκατάσταση της ε, φυσικής τάξης» και στην φυσική τάξη, αυτό το οποίο θέλει ο κύριος Βόιτ και ο κύριος Γιούρεκ, ε, υπάρχουν οι λευκοί straight χριστιανοί που επιβάλλουν τις αξίες τους και δεν δίνουν δικαιώματα σε άλλους. Γιατί δεν είστε ειλικρινείς. Και μιλήσατε για το μόνιμο πραξικόπημα και ανθρώπους που δεν οροδούν προουδενός. Μα μιλούσατε για τον εαυτό σας όμως τότε. Αυτή είναι η πραγματική σας ε, ατζέντα. Θα ήθελα λοιπόν να πω το εξής. Πρώτα απ' όλα, όπως ξέρετε υποστηρίζω πλήρως όλες τις ε, παρεμβάσεις ε, που κάνετε σε σχέση με την πολωνική κυβέρνηση η οποία έχει εξτρεμιστικές απόψεις. Το θέμα δεν αφορά τον πολωνικό λαό και μάλιστα οι μαζικές διαδηλώσεις στην Πολωνία ήταν υπέρ των αξιών που εκπροσωπούμε εδώ πέρα οι περισσότεροι. Αλλά κάτι το οποίο έχω επανειλημμένα υπογραμμίσει είναι ότι θεωρώ πως με το να εστιάζουμε συνεχώς στην ε, δικαιοσύνη ε, δεν ε, ωφελούμε τους εαυτούς μας. Πρέπει να δούμε ακριβώς το συστημική φύση του προβλήματος και τα είπε και η κυρία Μαλιμπιόρκ και έχουμε απευθύνει και μία επιστολή. Ακριβώς αυτό το οποίο λένε, δηλαδή να απαγορευτεί τελείως η έκτρωση, οι περιορισμοί στο δικαίωμα του συνέρχεστε, αλλά και η άρνηση να αναγνωριστεί η εξουσία του 10 και το πώς χρησιμοποιούνται οι λεγόμενες μεταρρυθμίσεις στην δικαιοσύνη για να προωθηθεί η ατζέντα την οποία μόλις ανέφερα. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να δούμε το πώς η πολιτική κυβέρνηση καταστρέφει την εξαρτησία της δικαιοσύνη, αλλά και όλα τα άλλα δικαιώματα και τις αξίες που κατά πλειοψηφία εδώ εκπροσωπούμε. Το θέμα λοιπόν δεν αφορά την Πολωνία και τον πολωνικό λαό. Είναι ακριβώς ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ως μια κοινότητα αξιών. Γι' αυτό ακριβώς προωθούμε αυτές τις αξίες και δεν ε, ε, μπορούμε να το βλέπουμε το ζήτημα καθαρά τεχνικά. Σας ευχαριστώ. Κυρία Ζνιεύσκα. Πάνε Panie Komisarzu, W μετά από τα προηγούμενα σχόλια, δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Διότι όλα αυτά είναι απόψει τη αντιπολίτευση που εκπροσωπείται εδώ. Συγγνώμη. Εγώ έχω εκλεγεί στην Πολωνία, είμαι υπερήφανη που είμαι Πολωνία εξελέγει για να υπερασπίζουμε την Πολωνία στην Ηνωμένη Ευρώπη και θέλω να πω στον Πρόεδρο ότι η κατάσταση έτσι όπως παρουσιάστηκε από τους προλαλήσαντες και που και αυτοί είναι εκλεγμένοι στην Πολωνία δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Κυρία Κουντρέτσκα, στην ομιλία της χρησιμοποίησε ε, απαράδεκτη γλώσσα. Μίλησε για προγραφές, μίλησε για έλεγχο, για κυδαιμονία. Αυτά τα πράγματα δεν ταιριάζουν στη σημερινή Πολωνία. Ευτυχώς δεν έχουμε αυτά που Είχαμε την προηγούμενη κυβέρνηση που παρακολουθήσαμε του δικαστέ, παρακολουθήσαμε τηλεφωνικέ συνδιαλέξει κλπ. Λοιπόν, η σημερινή κατάσταση στην Πολωνία είναι μια χαρά. Και το λέω αυτό διότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πέρσι είχαμε δηλώσει όσον αφορά την πορεία τη ανεξαρτησία. Πολωνοί πατριώτε έγιναν αντικείμενο προσβολών για τα 100 χρόνια λοιπόν τη ανεξαρτησία, 150.000 άνθρωποι παρέλεσαν στο κέντρο τη Βαρσοβία. Και σε πολλέ άλλε πόλει, στα χωριά, παντού. Ο κόσμο γιόρτασε τα 100 χρόνια τη πολωνική ανεξαρτησία. Μια χαρά λοιπόν είναι η κατάσταση στην Πολωνία. Και αυτό ισχύει και για την μεταρρύθμιση τη δικαιοσύνης. Ελπίζω να δείτε τι με το πράγμα και να λάβετε σοβαρά υπόψη τι απαντήσει που έδωσαν οι πολωνικέ αρχέ στην Κομισιόν και να παραδεχτείτε ότι οι αλλαγέ που γίνονται οδηγούν την Πολωνία στη σωστή κατεύθυνση. Ιδιαίτερα όσον αφορά τη μεταβολή του ορίου συνταξιδότηση από τα 70 στα 65. Ίσα ίσα, προηγούμενε κυβερνήσει αύξησαν το όριο κατά 12 χρόνια, το οποίο ήταν προσβολή για τους Πολωνούς και τις Πολωνέζες. Εμείς λοιπόν υπερμηνόμεθα του δικαιώματος ελεύθερης επιλογής των δικαστών όταν συνταξιοδοτούνται. Πρόεδρος, κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την υπομονή σας. Ε, μίλησαν πολλοί βουλευτές. Δεν ξέρω αν έχετε λίγο χρόνο να πείτε δύο λόγια, να απαντήσετε. Δεν είχαμε τόσο ερωτήσει όσο σχόλιο, οπότε αν νομίζετε έχετε τον λόγο. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στα όσα ακούστηκαν και να απαντήσω ενδεχομένω και κάποιε από τις ερωτήσεις που τέθηκαν. Θα σας πω πρώτα απ' όλα ποια είναι η πηγή της αισιοδοξία μου. Είναι ο ίδιος ο πολωνικός λαός. Η κοινωνία των πολιτών είναι ζωντανή, είναι δραστήρια. Οι Πολωνοί σκέπτονται ανεξάρτητα και ξέρετε, χωρί αυτού, ό,τι και να κάνουμε εμεί, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεν θα έχει και καμία ουσία. Όμω, χάρη στον πολωνικό λαό, στο τέλο θα πετύχουμε. Διότι, εν τέλει, η συντριπτική πλειονότητα του πολωνικού λαού θέλει να ανήκει σε αυτήν την κοινότητα πολιτών που ονομάζεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συντριπτική πλειονότητα. Ορισμένοι με επέκριναν τα τελευταία τέσσερα χρόνια, λέγοντας «Πρόσεξε γιατί αυτά που κάνεις θα γεννήσουν πάρα πολλούς ευρωσκεπτικιστές στην Πολωνία. Θα φύγει μακριά η Πολωνία από την Ευρωπαϊκή Ένωση». Και όμως το αντίθετο ακριβώ έγινε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πιο δημοφιλή στην Πολωνία. Οι Πολωνοί λοιπόν δεν χρειάζονται υποδείξει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται και σκέφτονται πολύ ευρωπαϊκά θα έλεγα. Το οποίο με οδηγεί στο δεύτερο πράγμα που ήθελα να πω στην πολωνική κυβέρνηση εν προκειμένου εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εάν θέλετε ο πολωνικό λαός να είναι μέρος αυτής της κοινότητα αξιών πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι κοινότητα αξιών σημαίνει και κανόνες που κάποιο πρέπει να σέβεται. Έχει πολλά ωφέλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά έχει και κανόνες. Και ένα από τους θεμελιώδεις κανόνες αυτής της λέσχης του πει, είναι το κράτος δικαίου. Αλλιώς δεν λειτουργούμε. Η κοινότητα αυτή δεν λειτουργεί. Και το λέω όχι μόνο ενώπιση των αρχών μα, αλλά και για πολύ πρακτικούς λόγου. Η εσωτερική μα αγορά λειτουργεί. Διότι κάθε πολίτης, κάθε επιχείρηση είναι βέβαιο ότι οι νόμοι τη Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο παντού. Μόνο έτσι λειτουργεί έχει, και έχει νόημα η ιστορική αγορά. Και ποιο ελέγχει κατά πόσον αυτό ισχύει ή όχι, οι εθνικοί δικαστέ. Υπάρχει την έννοια και με αυτή την ιδιότητα ο εθνικό δικαστή είναι ευρωπαϊο δικαστή. Εάν ο εθνικό δικαστή έχει κάποιε αμφιβολίε όσον αφορά την ορθή εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας στη χώρα του, μπορεί να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να ζητήσει συμβουλή για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Και προκειμένου με αυτήν την έννοια και πάλι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι εθνικό δικαστήριο. Και αυτός είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις χώρες, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό που περιέγραψα πρέπει να μπορεί να το κάνει ο εθνικό δικαστή ανεξάρτητα. Αν κάποιος λοιπόν τον εμποδίσει στη διαδικασία αυτή, τότε παρεμποδίζεται και η εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου. Ευθέως. Ευχαριστώ λοιπόν την προσοχή σα σε αυτό ακριβώ το γεγονό. Πρόκειται για κάτι το οποίο είναι απολύτω απαραίτητο για την ίδια τη λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα δικαστήρια δηλαδή είναι ανεξάρτητα και οι δικαστέ είναι όχι μόνο επαγγελματίε αλλά και ανεξάρτητοι στην εφαρμογή του νοσιακού δικαίου στι χώρε μέλη. Και επιτρέψτε μου και μια δεύτερη παρατήρηση. Ναι, ξέρω ότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε σήμερα, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα τη ακρόαση. Θα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Εν γένει όμω, οφείλω να πω το εξή. Η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και το κράτο δικαίου είναι κάτι το οποίο αφορά και τον τελευταίο πολίτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί κάθε πολίτη, άνδρα ή γυναίκα, πρέπει να νιώθει προστατευμένο από τον νόμο, όπω κάθε άλλο, χωρί διακρίσει. Αυτό είναι το θεμελιώδες στοιχείο, είναι ο πυρήνας του κράτους δικαίου. Δεν επιτρέπονται λοιπόν διακρίσει ει βάρο μια μειονότητα ή βάση του χρώματο του δέρματο ή τη θρησκεία κ.ο.κ. Ο νόμο δεν μπορεί να είναι το όργανο της πλειοψηφία για να ελέγξει την μειοψηφία για το τι κάνει και τι είναι. Αυτό έχει θεμελιώδη σημασία για το ποιοι είμαστε και πώς λειτουργούμε. Και γι' αυτό όλα αυτά είναι θεμελιώδες στοιχείο της δημοκρατίας μας. Γι' αυτό πρέπει να προστατεύσουμε την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, να προστατεύσουμε το κράτος δικαίου και τους κανόνες δικαίου. Σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που χαρακτηρίζεται από διαφορετικότητα, που όμως υπάρχει κάτι κοινό, ότι όλοι την χάνουν προστασία από τον νόμο. Είμαστε λοιπόν μια Ευρωπαϊκή Ένωση με πολλέ μειονότητε. Αν το καλοσκεφτείτε, ακόμα και η μεγαλύτερη χώρα, η Γερμανία, είναι μια μειονότητα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό, για άλλο ένα λόγο λοιπόν, χρειαζόμαστε τον, το κράτο δικαίου για να μην δεσπόζει ποτέ, να μην επικρατεί ποτέ ολοκληρωτικά μια πλειονότητα, μια πλειοψηφία. Αυτό συζητούμε λοιπόν εδώ σήμερα. Και αυτό. Διότι ποιοι θα ήταν τα πρώτα θύματα εάν δεν ίσχυε το κράτο δικαίου. Οι μειονότητε. Από αυτού ξεκινάμε πάντα. Αυτοί είναι τα πρώτα θύματα πάντοτε. Και δεν είναι τυχαίο που πολλέ μειονότητε βρίσκονται υπό τέτοια τεράστια πίεση στι μέρες μας στην Ευρώπη. Αυτές λοιπόν θα ήταν οι επιπτώσει. Όπω είπα, άγνοια του κρατούς δικαίου θα οδηγούσε σε κατακαιρματισμό της Ευρωπαϊκής Ένωση. Αν οι Πολωνοί θέλουν να παραμείνουν μέρος αυτής της κοινότητας αξιών, τότε αυτές οι αξίες πρέπει να τύχουν προστασίες Και αυτό είναι καθήκον κάθε αρχής, κάθε εθνικής αρχής. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βεβαίως είναι ο θεματοφύλακας αυτών των υποχρεώσεων. Και παρεμβαίνουμε κάθε φορά που βλέπουμε να απειλούνται. Ο κ. Γιούρεκ μίλησε για τα πολωνικά δικαιώματα. Σας είπα τι πιστεύω. Διαφωνώ λοιπόν, αλλά αυτή είναι η επίσημη θέση της Κομισιόν και θα του λέω το εξή. Κάτι είπε για την άρνηση έκδοση. Αυτό οι δικαστές μπορούν να το πράξουν, αν δηλαδή στον Ευρωπαϊκό Δικαστικό Χώρο, που είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο, εάν κάποιο θέλει να ζητήσει την έκδοση, κάποιο από κάποια άλλη χώρα, εκεί έχουμε έναν δικαστή, ο οποίος πρέπει να είναι σίγουρος ότι αυτό που αντιμετωπίζει δίωξη σε κάποια άλλη χώρα θα αντιμετωπίσει εκεί μια δίκαιη δίκη. Και λυπούμε, αλλά εδώ έχουμε αμφιβολίες περί αυτού. Λόγω ακριβώ του σορευτικού αποτελέσματο αυτών που συμβαίνουν στην Πολωνία, στη δικαιοσύνη, στην εκτελεστική εξουσία κλπ. Κάποιοι δικαστέ, λοιπόν, έχουν αμφιβολίε. Τα αποφασίσει το δικαστήριο ή θα αποφασίσει μετά από κάποιο τηλεφώνημα από τον Υπουργό. Εκεί βρισκόμαστε δυστυχώ σήμερα. Και μόνο τρόπο να τα σταματήσουμε όλα αυτά. Να επιτρέψουμε λοιπόν να δικάζουν οι εγκληματίε πρέπει ε, προποθέτει ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Θα προσφέρετε κύριε Γιούρα και υπηρεσίε στον πολωνικό λαό αν φροντίζετε η πολωνική δικαιοσύνη να είναι ανεξάρτητη. Έτσι οι εγκληματίε θα καταλήξουν στη φυλακή. Γι' αυτό και, ε, ξέρετε, στην υπόλοιπη Ευρώπη οι δικαστέ δεν έχουν κανένα πρόβλημα να στείλουν, να εκδώσουν κάποιο ή κάποια άλλη χώρα, γιατί έχουν πρόβλημα με την Πολωνία. Κύριε Ιρεκ, εγώ προσωπικώ είμαι αρμόδιο στην Κομισιόν για το άρθρο 17 και παρόμοιου διαλόγου έχουμε τακτικά με εκπροσώπους της Πολωνίας, με εκπροσώπου τη Πολωνική Καθολική Εκκλησία. ή την Ρωμαϊκή, καθολική, τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία της Πολωνίας, αν θέλετε. Και πρέπει να σας πω ότι οι εκπρόσωποι της Εκκλησίας με τους οποίους μίλησα αναφέρονται όλοι τους στο δόγμα που λέει ότι πρέπει να σέβεσαι το Σύνταγμα, να ξέρετε ότι είναι δόγμα της Ρωμαιοκαθολική Εκκλησίας στην Πολωνία. Ναι. να ξέρετε και η Εκκλησία είναι μέρος του διαλόγου για την κοινωνία των πολιτών και τα δικαιώματα. Και το κάνουμε αυτό με όλες τις εκκλησίες ανά την Ευρώπη, ε, αλλά και με μη θρησκευτικού χαρακτήρα οργανώσεις. Κάνουμε μεγάλη προσπάθεια, να το ξέρετε. Και κάνουμε, κάνουμε πολλή προσπάθεια τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Το κάνουμε και με την ε, Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία της Πολωνίας. Αυτό το λέω για να είμαστε εντελώ ξεκαθαροί. Και να κλείσω λέγοντα το εξή, που είναι πολύ σημαντικό για μένα έχουμε μια τελείως διαφορετική όψη της κοινωνίας. Δεν συμμερίζομαι τον στενό ορισμό του χριστιανού που υιοθέτησε ο κ. Βόκτ. Ούτε συμμερίζομαι τον βαθύ θαυμασμό του κύριου Βόκτ για τον Πούτιν. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω προς τους πολλούς φίλους είναι προσέχετε ποιοι σας κολακεύουν, ποιοι σας επικρίνουν και ποιοι σας επιβραβεύουν. Αυτά ευχαριστώ. Thank you uh, Ευχαριστούμε πολύ, Επίτροπε. Οπότε τώρα ολοκληρώσαμε και σας ευχαριστούμε για το χρόνο σας, τις απαντήσεις. Συνάδελφοι, πριν προχωρήσουμε στο επόμενο πάνελ που αφορά τα θεσμικά όργανα Επαναλαμβάνουμε ότι πρόκειται για μια διαδικασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Κοινοβούλιο ε, έχει συνενέσει. Και οπότε τώρα έχουμε κάποιες πάρα πολύ σύντομες ε, δηλώσεις από την Αυστριακή και την Ρωμανική Προεδρία για να ενημερωθούμε όσον αφορά την σχετική διαδικασία και πώς προχωράει. Πρώτα-πρώτα έχουμε τον ε, νομικό σύμβουλο της ε, μόνιμης αντιπροσωπής της Αυστρίας και θα μας ενημερώσει για τα θέματα αυτά που συζητούμε, το τι θα γίνει κατά την Αυστριακή Προεδρία. Έχετε τον λόγο. Κύριε Πίτνερ, έχετε τον λόγο. Μπίτνερ. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι βουλευτές, είναι θεμελιώδη αξία τη Ένωση Το κράτος δικαίου και η ανεξάρτητη δικαιοσύνη είναι το κλειδί για την λειτουργία της ενιαία αγοράς και για να λειτουργεί και η δικαστική συνεργασία. Από το 1917 το Σεπτέμβριο ενεργοποίησαμε το άρθρο 7 κατά της Πολωνίας. Για πρώτη φορά επικαλεστήκε η Ένωση αυτή τη διαδικασία. Να σας ενημερώσω τι έγινε από τότε στο Συμβούλιο. Η πρώτη ευκαιρία για να ε, ασχοληθούμε με το άρθρο 7 αφού το ενεργοποιήθηκε ήταν το Συμβούλιο Γενικοπαίδων 27 Φεβρουαρίου οπότε τότε ενημερώθηκαν οι Υπουργοί για το πώς έχουν τα πράγματα και συγκεκριμένα για τον συνεχή διάλογο με την Πολωνία με σκοπό την εξέβρεση κάποιες λύσεις. Ε, μετά, σε άλλη συνάντηση του Υπουργείου Νοικοπαθήσεων, στις 23 στις 17 Απριλίου και 14 Πέμπτου ενημερώθηκαν οι Υπουργοί για τις εξελίξεις στην Πολωνία. Οι Υπουργοί είπαν ότι συμφωνούν να συνεχιστεί ο διάλογος. Και στα πλαίσια του διαλόγου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Πολωνία τροποποίησε την ομοθεσία της. Παρ' όλα αυτά η Επιτροπή θεώρησε ότι αυτά δεν αρκούν και έτσι δεν καλύπτονται οι βασικές ανησυχίες. γι' αυτό ζητήθηκε επίσημη ακρόαση για να γίνει ε, με την Πολωνία. Αυτό έγινε στις 26 έκτου στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων και έτσι ενημερώθηκαν οι Υπουργοί για τα όσα ε, αποτέσαν τα ελαττήρια αυτής της πρότασης. Οπότε για να κατοχυρωθούν τα οικονομικά διαδικαστικά δικαιώματα της Πολωνίας ε, αποφασίστηκαν κάποιες διαδικασίες στις 18 δε Σεπτεμβρίου έγινε μια δεύτερη τέτοια συνάντηση, μια δεύτερη ακρόαση με την ίδια διαδικασία όπως είχε γίνει και στην ακρόαση της 26ης Ιουνίου. Συνεχίστηκε και εις βάθος η ανταλλαγή των απόψεων με τους υπουργούς και την χώρα. Ε, βασικά για τα θέματα της εξαρτησίας της δικαιοσύνης και των ε, εγγυήσεων ότι τηρούνται αρχές του κρατού δικαίου στην ασκή τη δικαιοσύνη. Στι 16 Δεκάτου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε για τι πρόσφατε εξελίξει για τη μεταρρύθμιση τη δικαιοσύνη. και παρέφεραν οι Υπουργοί το ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το να ισχύει το κράτο δικαίου σε όλα τα κράτη-μέλη και τόνισαν ότι θα πρέπει να υπάρξει χειροπιαστή πρόοδο Τον Νοέμβριο Επίσης η Επιτροπή ενημέρωσε τους Υπουργούς και τώρα για το τελευταίο ε, συμβουλευτικών υποθέσεων. Η Προεδρία μας θα ενημερώσει και θα ξαναβάλει στην διάταξη το άρθρο για την Πολωνία. Εμείς παίρνουμε στα σοβαρά την υπόθεση αυτή και για αυτό ε, προκαλούμε με κάθε σεβαθμό της διαδικασίας του άρθρου την ε, συζήτηση στο Συμβούλιο. Πάντως ελπίζουμε ότι ο διάλογος μεταξύ της Κομισιόν και της χώρας θα αποδώσει καρπούς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εμείς ευχαριστούμε κύριε Μπίτνερ. Και, ε, θα ε, ακούσουμε και την ε, Ρουμανική Προεδρία των Ρουμάνο μόνιμο εκπρόσωπο καθώς η Ρουμανική Προεδρία είναι η επόμενη να μας πει πώς θα αντιμετωπίσει το ζήτημα κατά τη διάρκεια της ε, Προεδρίας της Ρουμανίας. Σύντομα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες ε, και κύριοι βουλευτές και αγαπητοί εκπρόσωποι του Συμβουλίου και της ε, Επιτροπής. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και για το ότι μας δώσετε την δυνατότητα να σας παρουσιάσουμε το πόσο βλέπουμε το άρθρο 7 και την διαδικασία αυτή Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω, να τονίσω τα όσα ακούστηκαν από τους προηγούμενους ομιλητές, ε, ότι δηλαδή το κράτος δικαίου είναι θεμελιώδης αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και αυτό είναι κάτι το αναμφισβήτητο. Εμείς θα ξεκινήσουμε με βάση τα επιτεύγματα της ε, προηγούμενης ε, Προεδρίας και ήδη ο Αυστριακός συνάδελφος σας είπε πώς έχουν τα πράγματα στο Συμβούλιο και παίρνουμε το θέμα πολύ στα σοβαρά, σεβόμενοι πλήρως τις ε, συνθήκες και θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο του άρθρου 7 μιλάμε για την λεγόμενη προληπτική διαδικασία στο πλαίσιο του κράτους δικαίου και γι' αυτό θεωρούμε ότι όλες ε, θα πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να υπάρχει επικοδομητικός διάλογος μεταξύ όλων των μερών και ως ε, διαμεσολαβητής θα διευκολύνουμε την διαδικασία και τον διάλογο και ελπίζουμε βεβαίω ε, τα μέρη του διαλόγου, η Κομισιόν και η Πολωνία δηλαδή, θα συνεχίσουν να έχουν επικοδομητικές ε, επαφές ε, κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τους δύο συναδέλφους από την Αυστριακή και την Ρουμανική Προεδρία. Περνάμε τώρα στο θεσμικό μας ε, πάνελ και θα ακούσουμε τώρα πρώτα απ' όλα τον επίτιμο Ζαν Κλωτ Σόλτσεν, τον κύριο Κίστερ και πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συμβουλίων Δικαιοσύνης και τον ε, δόκτωρα Άνταμ Μπόντναρ, τον ε, Πολωνό συνηγόρο του πολίτη. Λοιπόν, έχετε 10 λεπτά ο καθένας. Έλατε εδώ μπροστά, πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η Επιτροπή της Βενετίας έχει ασχοληθεί εντατικά με το φάκελο Πολωνία κατά τη διάρκεια των ετών 2016 και 2017. Το μικρόφωνο του ομιλητή δυστυχώς είναι κλειστό ως ένα εκ των παλαιότερων μελών της Επιτροπής αυτής. Δεν έχω δει άλλο φάκελο τόσο δύσκολο από όλες τις απόψεις. Θα μιλήσω για δύο αλλαγέ που έγιναν στην Πολωνία. Δύο γνώμες εξεδόθηκαν το Δεκέμβριο του 2017. Η μία αφορά τη Γενική Εισαγγελία. Ο δεύτερος ε, αφορά το Εθνικό Συμβούλιο Δικαιοσύνη, την οργάνωση του Ανατολικού Δικαστηρίου και των τακτικών δικαστηρίων. Η έναρξη των εχθροπραξιών, ούτως υπήν, ε, έγινε με αφορμή το συνταγματικό δικαστήριο και για να κατανοήσει κανείς την κατάσταση πρέπει να πάμε πίσω στην περίοδο πριν από την ε, ανάληψη της εξουσίας το 2015 από το κόμμα Νόμος και Δικαιοσύνη. Την εποχή εκείνη η κυβέρνηση είχε ε, κυριαρχό κόμμα, την πλατφόρμα των πολιτών και τότε ψηφίστηκε μια τροποποίηση, μια τροπολογία η οποία έδινε το δικαίωμα στην κατοβουλή να εκλέγει τους δικαστές και συγκεκριμένα αυτούς οι οποίοι θα το κατά τη διάρκεια του 2015. Οι τρεις εν προκειμένου θα έπρεπε να γίνουν αντικείμενο διαδοχή, οι δύο όμω θα συνέχιζαν και θα επελέγονταν από την επόμενη Βουλή. Αυτό είχε αποφασίσει το Συνταγματικό Δικαστήριο με αποφάσεις του τον Δεκέμβριο του 2015. Οι αποφάσεις αυτές δεν εφαρμόστηκαν ποτέ από τις πολωνικές αρχές. Οι τρεις δικαστές που είχαν κανονικώς εκλεγεί σύμφωνα με την εντολή του Συνταγματικού Δικαστηρίου ποτέ δεν έδωσαν τον όρκο τους ενώπιον του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Αντιθέτως, το νέο κοινοβούλιο όρισε πέντε νέους δικαστές, δύο συμφώνως με την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, οι τρεις όμως ορίστηκαν κατά παράβαση της εν λόγω απόφασης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, μάλιστα, όκησε αμέσως χωρίς την παραμικρή καθυστέρηση και τους πέντε αυτούς δικαστές. Οι πολωνικές αρχές περίμεναν με ανυπομονησία την εκπνοή της εντολής του Πρόεδρου του Δικαστηρίου, του κ. Αντρές Στι στις 19 Δεκεμβρίου του 2016. Την εποχή εκείνη, τη στιγμή εκείνη, ψηφίστηκαν ε, φωτογραφικοί νόμοι. Ορίστηκε νέα πρόεδρος υπό συνθήκες πραγματικές και νομικές, μάλλον αμφίβολες και μάλιστα η πρώτη πράξη της νέας πρόεδρου ήταν να δεχθεί να δικάσουν οι τρεις δικαστές οι οποίοι είχαν οριστεί με τρόπο αντισυνταγματικό. Η κατάσταση αυτή επιβιώνει ως και σήμερα και βεβαίως είναι μια κατάσταση η οποία πλήττει την αξιοπιστία του συνταγματικού δικαστηρίου, του οποίου η ίδια η σύνθεση είναι αντισυνταγματική. Πέραν αυτών των προβλημάτων που αφορούν τη σύνθεση την ίδια του συνταγματικού δικαστηρίου, και άλλε τροπολογίε έπληξαν την ίδια τη λειτουργία του. Αυτό που θα μπορούσε να πει κανεί για αυτέ τι τροπολογίε είναι ότι είχαν ένα σαφή στόχο να επιβραδύνουν, αν όχι να παρεμποδίσουν ολοκληρωτικά, τη λειτουργία του δικαστηρίου. Για να σα δώσω ένα μόνο παράδειγμα, η ολομέλεια του δικαστηρίου μπορεί να αποφασίσει με παρουσία 13 εκ των 15 δικαστών και με πλειοψηφία 2 τρίτων Εν προκειμένου, οι επικρίσεις της Επιτροπής της Βενετίας τον Μάρτιο του 2016 ήταν εντονότατε. Μάλιστα, εντωμεταξύ, το Συνταγματικό Δικαστήριο ακύρωσε αυτέ τι τροπολογίε. Παρόλα αυτά, η κυβέρνηση αρνήθηκε να δημοσιεύσει τη σχετική απόφαση, όπω και άλλε αποφάσει εν συνεχεία, παρά το γεγονό ότι το ίδιο το Σύνταγμα επιβάλλει άμεση δημοσίευση των αποφάσεων του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Η δεύτερη γνώμη της Επιτροπής της Βενετίας επί του Συνταγματικού Δικαστηρίου συζητήθηκε στην συνεδρίαση του Οκτωβρίου του 2016. Η υπόθεση αυτή ξεκίνησε ε, με πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης και αφορούσε την νιωστή τροπολογία, ε, τροποποίηση μάλλον του νόμου για το Συνταγματικό Δικαστήριο. Ήθιστε στην Επιτροπή της Βενετίας να παρίσταται η χώρα αντικείμενο της συζήτησης. Παρ' όλα αυτά οι πολωνικές αρχές αρνήθηκαν να εμφανιστούν. Εν πάση περιπτώσει, εν τω μεταξύ κάποιες ε, ακραίες κινήσεις διορθώθηκαν, όμως παραμένει γεγονός ότι η βασική πρόθεση των πολωνικών αρχών ήταν να κερδίσουν χρόνο προτιμάζοντας την εξ ολοκλήρου και δαιμόνευση του ανωτάτου δικαστηρίου. Περιμένοντας δηλαδή την αποχώρηση του πρώην Προέδρου του δικαστηρίου τον Δεκέμβριο του 2016 όπως ε, προανέφερα. Έκτοτε το συνταγματικό δικαστήριο έπεσε θύμα συρρήκνωσης της φήμης του, της αξιοπιστία του. Μάλιστα πολλές προσφυγές αποσύρθηκαν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το αναφέρει κανείς, διότι Πολλοί νόμοι δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν ως προς την εφαρμογή τους χωρίς προσφυγή στο συνταγματικό δικαστήριο. Έτσι, το συνταγματικό δικαστήριο γίνεται όλο και περισσότερο ένα απλό δικονομικό όργανο στα χέρια της κυβέρνησης, η οποία το αξιοποιεί όπου τη βολεύει. Όσον αφορά τα της δικαιοσύνης γενικότερα, αξίζει να υπενθυμίσουμε τον νόμο για την Γενική Εισαγγελία, τον οποίο σχολίασε η Επιτροπή της Βενετίας τον Δεκέμβριο του 2017. Δεν υπάρχει εμβολία, γεγονός ότι η Γενική Εισαγγελία μπορεί να οργανωθεί με διαφορετικούς τρόπους σε κάθε χώρα δεν μπορούμε εδώ να μιλάμε για τους εισαγγελείς όπως για τους δικαστές. Όμως και εδώ βλέπουμε ότι η πολωνική κυβέρνηση προσπάθησε να συμπήξει 100% τον ρόλο του Υπουργού Δικαιοσύνη με τον ρόλο του Γενικού Εισαγγελέα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να συγχαίεται η διάκριση των εξουσιών. Το Δεκέμβριο και πάλι του 2017 ψηφίστηκαν άλλοι τρεις νόμοι για τους οποίους εξέδωσε γνώμη η Επιτροπή της Βενετίας. Αφορούν το Ανώτερο Συμβούλιο της Δικαιοσύνης, το Ανώτερο Δικαστήριο και άλλα δικαστήρια. Όσον αφορά το Ανώτερο Συμβούλιο Δικαιοσύνης, το οποίο εκ του συντάγματος έχει το καθήκον να εγγυάται την ανεξαρτησία των δικαστικών. Σύμφωνα λοιπόν με αυτόν τον νόμο, τα 15 μέλη που εκπροσωπούν τους δικαστές δεν εκλέγονται από τους ίδιους τους δικαστές, αλλά από την κάτω βουλή. Κάτι το οποίο γύρει κίνδυνο βεβαίως πολιτικών επιλογών. Επιπλέον, όλα τα μέλη του σημερινού Συμβουλίου Δικαιοσύνης εκπαραθυρώθηκαν και θα αντικατασταθούν. Επίσης, το ανώτερο δικαστήριο. Και αυτό μεταρρυθμίζεται εκ βάθρων. Δημιουργήθηκαν δύο σώματα. Το ένα είναι πειθαρχικού χαρακτήρα και το άλλο δέχεται κάτι καινοφανέ, εξαιρετικές προσφυγές, έκτακτες προσφυγές. Έχει μάλιστα το δικαίωμα αυτό το δεύτερο σώμα να επανεξετάζει κάθε δικαστική απόφαση των τελευταίων 20 ετών. Κάτι το οποίο πλήττει βεβαίω και την κοινωνική δικαιοσύνη και το κράτο δικαίου. Αυτά όλα μα θυμίζουν δυστυχώ το παλαιποτέ σοβιετικό σύστημα. Τον αμφισβητεί κανεί εκ βάθρων όλε τι αποφάσει, όλε τι δικαστικέ αποφάσει τη τελευταία 20 ετία, κάθε άλλο παρά υπηρετεί την ασφαλή δικαίου. Και ω προ το Ανατολικό Δικαστήριο, εδώ μειώθηκε το όριο συνταξιοδότηση αμέσω από τα 70 στα 65 έτη. Κάτι το οποίο αφορά περίπου ένα τρίτο των ε, σημερινών δικαστών, κάτι το οποίο αποσκοπεί στη δημιουργία νέων θέσεων που θα πληρώσει η σημερινή κυβέρνηση. Μάλιστα κάποιοι δικαστές και από ό,τι φαίνεται αυτοί οι συγκεκριμένοι δικαστές θα έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν από τον ε, πρόεδρο της, της Δημοκρατίας να παρατείνει την ε, εντολή τους, τη θητεία τους. Τέλος, όσον αφορά τα τακτικά δικαστήρια, οι πρόεδροι των δικαστηρίων όλων των επιπέδων έχουν σημαντικές εξουσίες και αρμοδιότητες. Όμως, το σύστημα, η πολωνική δικαιοσύνη είναι οργανωμένη με εξαιρετικά ιεραρχικό τρόπο. Οι πρόεδροι των κρατέρων δικαστηρίων είναι υπεύθυνοι και αναφέρονται στους πρόεδρους των μεσαίων και ανωτέρων δικαστηρίων και αυτοί απευθεία στον Υπουργό Δικαιοσύνη. Ο τελευταίος μπορεί να ανακαλέσει πρόεδρους δικαστηρίων, κατά το οποίο μπορεί να ανατραπεί μόνο από το Ανώτερο Συμβούλιο Δικαιοσύνης, το οποίο όμως πλέον είναι ένα πολιτικό όργανο και το οποίο αποφασίζει με πλειοψηφία δύο τρίτων, κάτι το οποίο είναι εντελώς πλέον αδύνατον. Και σε κάθε περίπτωση έχουμε και μεταβατικέ διατάξει, οι οποίε ενισχύουν ακόμη περισσότερο τι αρμοδιότητε του Υπουργού Δικαιοσύνη. Όπω προείπα λοιπόν, ε, ο Υπουργό Δικαιοσύνη είναι πλέον και Γενικό Εγγελέα, κάτι το οποίο αυξάνει υπέρμετρα, εκθετικά θα έλεγα, την επικυριαρχία του επί τη δικαιοσύνη. Εν κατακλείδη και συνοψίζοντα, δεν έχουμε πλέον συνταγματικό έλεγχο. Ο Υπουργό Δικαιοσύνη ταυτίζεται πλέον με τον Γενικό Εισαγγελέα, κάτι το οποίο αντιβαίνει στη γενικότερη τάση στην Ευρώπη, ε, που κατατείνει στην εξαρτησία της Γενικής Εισαγγελίας και η δαιμόνευση του Ανωτάτου Συμβουλίου Δικαιοσύνης. Οι δικαστές εκλέγονται πλέον από την Κατοβούλη. Το Ανώτερο Δικαστήριο μπορεί να ανατρέψει τις αποφάσεις των τελευταίων 20 ετών μείωση, άμεση μείωση της ηλικία συνταξιοδότησης των δικαστών του Ανώτατου Δικαστηρίου. Ε, μάλιστα υπάρχει μια επιβαρυντική <laughs> περίσταση. Οι νέοι δικαστές έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν παράταση της θητείας τους κατά εξαίρεση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και τέλος, πολύ σημαντικές πιέσεις επί των Προέδρων των δικαστηρίων όλων των επιπέδων ε, στο πλαίσιο μιας δικαιοσύνης που έχει πυραμιδοειδή ε, δομή με επικυρίαρχο των πάντων εν τέλει και κριτή των πάντων τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Κυρίε και κύριοι, ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Εμείς ευχαριστούμε καθηγητά Σόλσαμ. Είναι πολύ σημαντική η γνώμη της Επιτροπής της Βενετίας. Οπότε τα όσα είπατε θα τα λάβουν και εγγράφους οι συνάδελφοι, ούτως ώστε να μπορούν να έχουν μια πλησότερη, πληρέστερη, συγγνώμη, άποψη. Μη σηκώνεστε, έχουμε ρωταπαντήσει και τώρα πάμε στον κύριο Στέρκα. Α ζητούν να, μαθούν, να, δουν, την αφίσα τη ε, εκδήλωση τη ακρόασή μα. Οι Πολωνοί συνάδελφοι θα γνωρίζουν αυτή την εικόνα. Είναι το άγαλμα που απεικονίζει την ε, δικαιοσύνη στο Γκντάνσκ. Ε, συνήθως είναι βαρετά τα πόστερ, οι αφήσεις για τις εκδηλώσεις, αλλά αυτό για τη σημερινή εκδήλωση είναι πολύ ωραία. Πάμε τώρα. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Δικαστικών Συμβουλίων. Πρόεδρος του δικτύου είναι ο κύριος Κέι Στέρκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Πρώτα να σας μιλήσω για τον ε, φορέα μας. 24 δικαστικά συμβουλία δικαστών έχουμε στην φορέα μας. Και σήμερα μας είναι η ανεξαρτησία της ε, δικαιοσύνης. Δεν ασχολούμαι επομένω με τους δικαστές ως ε, άτομα, αλλά με τον φορέα της δικαιοσύνης. Και από τη μία μεριά έχουμε τη δικαιοσύνη και από την άλλη καλλιεστική εξουσία και εμείς είμαστε στην μέση ως ε, ουδέτεροι. Το 2018 αποφασίστηκε να ανασταλεί η συμμετοχή του Πολωνικού Συμβουλίου. Να σας πω τι ε, διαδικασία ακολούθησε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Όπως οι περισσότεροι θα γνωρίζετε, από τον ε, Οκτώβριο του 2015 το κόμμα της ε, δικαιοσύνης και του νόμου με τα ρυθμιστική. Από τότε, από το 2015, πρότεινε κάποιες αλλαγές και θέσπισε κάποιους νέους νόμους μεταξύ άλλων το πολιτικό το, το κοινοβούλιο άλλαξε τα σχετικά με το, το δικαστήριο, το Ισλαμικό Δικαστήριο, τα τακτικά δικαστήρια και το Δικαστικό Συμβούλιο και οι άρες. Θα έπρεπε οι δικαστέ να συμμετέχουν σε κάθε τέτοια μεταρρύθμιση, ούτω ώστε να εξασφαλιστεί η ανεξαρτησία δικαστική ουσία και επομένω έτσι να υπάρχει εμπιστοσύνη σε αυτέ τι μεταρρυθμίσει λοιπόν, και να είναι ισχυρές Όμω δεν είναι τίποτα τέτοιο. Δεν ρωτήθηκαν δικαστέ πάντοτε προσφέρουν τους δικαστές κάποια νομοσχέδια που δεν θα μπορούσε να αλλάξει κανένας. Οπότε επανειλημμένα οι δικαστές προέβησαν σε δηλώσεις και το δικαστήριο είπε ότι ανησυχεί για το μέλλον του Δικαστικού Συμβουλίου και ανησυχούσαμε ότι δεν πρόκειται να τηρείται ο κανόνας ότι θα πρέπει να είναι η δικαιοσύνη ανεξάρτητη με εξουσία κατά το οποίο αποτελεί κοινοτικό δίκαιο. Δεν ε, αντέδρασαν οι Πολωνοί, ούτε έγινε κανένας διάλογος. Η κυβέρνηση πράτησε επιφυλάξεις ε, του φορέα μας προχώρησε στη θέση αυτών των νόμων. Μετά τη θέση σε ισχύ του νόμου του Ιανουαρίου του 2016 είπαμε ότι δεν μπορεί να είπε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν μπορεί να συμμετέχει ε, ε, το Δικαστικό Συμβούλιο στο δικτυό μας τον Ιούνιο ε, επισκεφθήκαμε τον, την, την Πολωνία είδαμε τον Πρόεδρο δικαιοσύνη και θέμη, ένα φορέας με τον οποίο ήρθαμε σε επαφή ε, ήρθαμε σε επαφή επίσης και με τον Δημοσιολευτή που κάθεται δίπλα μου. Το Διευθυντικό Συμβούλιο απάντησε ε, στα όσα ε, είπε το δίκτυό μας και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Πριν σας πω κάτι για την ουσία, θα πρέπει να πω ότι όλοι στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο φάσουν τη λύπη τους για το θέμα αυτό εις βάρος του ε, Συμβουλίου Δικαστών της Πολωνίας που είναι ιδρυτικό μέλος του δικτύου μας αξιοσέβαστο και βοήθησε πάρα πολύ εδώ και πολλά χρόνια. Τώρα, πρώτα πρώτα, τι λέει το δικτύο μας, ότι θα πρέπει να εξετάσουν τι ισχύει για τους πολλού δικαστές και τόσα ισχύουν για το Ανώτο Δικαστήριο, το ευθυματικό Δικαστήριο και είναι σαφέ για το δικτυό μα ότι τώρα η εξουσία η, πέρασε από τους δικαστές στην ε, κυβέρνηση και επομένως ε, έχει γίνει παραβίαση τη ε, εξάρτητης δικαιοσύνης ή της αρχής ανεξάρτητη δικαιοσύνης και τα όσα είπε η κυβέρνηση δεν δικαιολογούν αυτήν την κατάργηση της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, οπότε θα σας πω μόνο τα σχετικά τα όσο διέπουν το Δικαστικό Συμβουλίο. Οι δικαστές πλέον δεν επιλέγονται από τους συναδέλφους τους, αλλά από το Κοινοβούλιο γίνεται ο διορισμός τους. και πρόκειται για τη συμμετοχή 2.000 πολιτών ή 25 δικαστών. Όμω εμεί λέμε ότι οι ομότιμοι θα πρέπει να του καλύπτουν και αυτό να κατά πλειοψηφία να γίνεται. Βέβαια, Εάν δεν ισχύει αυτό ο κανόνα, αυτό δεν σημαίνει ότι οι δικαστέ είναι ανεξάρτητοι από την κυβέρνηση. Αλλά στην περίπτωση των Πολωνών δικαστών υπάρχουν και άλλε μεταβλητέ. Μα οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι το Δικαστικό Συμβούλιο πλέον δεν έχει ανεξαρτησία. Τα εξή λάμπη υπόψη μα. Το σύνολο των νόμων αυτή τη μεταρρύθμιση για τον έλεγχο τη δικαστική εξουσία από την κυβέρνηση. Ο σκοπό ήταν υποτίθεται να είναι πιο αποτελεσματικό ο νόμο, να μην επηρεάζουν οι κομμουνιστέ, να υπάρχει ε, αποτελεσματικότητα. Παρ' όλα αυτά, το νέο Συμβούλιο και η κυβέρνηση δεν μα ξεκαθάρισαν πώ αυτέ οι μεταρρυθμίσει ακριβώ θα οδηγήσουν σε επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων. Και η διαδικασία επιλογής ενό μέλου του, του Συμβουλίου του δικαστικού δεν είναι κάτι που έχει διαφάνεια, δεν μπορεί κανείς να ελέγξει τα κριτήρια ε, και τι γίνεται με τους δικαστικούς που υπηρετούν στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ε, και για κάθε ότι έχουμε 25 ε, δικαστές ούτε ε, το Διαρκό Συμβούλιο μας είπε ποιοι είναι οι δικαστές που λαμβάνουν αυτή την απόφαση για την μεταρρύθμιση ούτε τα κριτήρια και οι περισσότεροι εξ αυτών είναι πάρα πολύ κοντά στην κυβέρνηση και στο κυβερνόν κόμμα. Τέσσερα από τα μέλη λίγο πριν εκλεγούν ως μέλη του Συμβουλίου ήταν αποσπασμένοι ως δικαστές στο Υπουργείο Δικαιοσύνη. Πέντε μέλη διορίστηκαν από τον Υπουργό Δικαιοσύνης μέσω της ειδική αρμοδιότητας που το απένιμε η μεταρρύθμιση. Και αυτός ο νόμος έγινε λίγο πριν ε, γίνει αυτός ο διορισμός και 14 από τους 25 είναι μέλη του Γευροντός Κόμματος ε, και τους ε, επέλεξε το Κοινοβούλιο κατόπιν προτάσεως της ε, κυβέρνησης και του κοινωνικού Κόμματος. Και έχουμε 10.000 δικαστές στην Πολωνία που θεωρούν ότι είναι πολιτικοποιημένοι οι δικαστές. Και τα μέλη του Συμβουλίου υποστηρίζουν όλες τις μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης. Οι περισσότεροι βέβαια των δικαστών θεωρούν ότι οι μεταρρυθμίσεις ε, είναι αντισυνταγματικές και ότι καταργούν την εξαρτησία της δικαιοσύνης. Πολλά μέρη του Δικαστικού Συμβουλίου είπαν ότι οι δικαστές που δηλώνουν πράγματα κατά της κατάρρευσης ανεξαρτησίας και κατά των μεταρρυθμίσεων θα πρέπει να απολυθούν με επιθαρικές διαδικασίες γιατί αυτό είναι παράνομη ε, δραστηριότητα. Επίσης, δεν λαμβάνει θέση υπέρ των δικαστών ε, το Δικαστικό Συμβούλιο όπως ε, ο πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Γι' αυτό το Σεπτέμβριο του 2018 σε έκτακτη συνεδρίαση 21 από τα 24 συμβούλια ε, ψήφισαν ε, να βγει από τον φορέα μας το Πολωνικό Συμβούλιο ένας, ένα, ένα συμβούλιο απέσχε και μόνο οι Πολωνοί ε, ψήφισαν κατά. Ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή η αποβολή από το δίκτυο των Πολωνών θα έρθει. Αλλά αυτό θα γίνει μόνο όταν οι αρχές που έχουν παραβιαστεί ξαναισχύσουν στην Πολωνία. Πάντως, δεν είμαστε αισιόδοξοι και μάθαμε ότι άρχισαν πληθυντικές διαδικασίες κατά των παλαιών μελών του Συμβουλίου, κατά των δικαστών που διαμαρτύρονται, κατά αυτών που ασκούν το δικαιωμά του ως Ευρωπαίοι δικαστές να στείλουν προδικαστικές ερωτήσεις στο δικαστήριο του Λουξεμβούργου. Θέλουμε να βελτιωθεί η συνεργασία, να υπάρξει αμοιβή κατανόηση μεταξύ των ε, δικαστικών συμβουλίων. Άρα θα πρέπει να υπάρξει κοινή ανάληψη ευθύνη για, την, ε, τις κοινέ αρχές που έχουμε και κυρίως όσον αφορά την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και το κράτος δικαίου. Τα κρατημένοι μπορούν να οργανώσουν τη δικαιοσύνη όπως νομίζουν ότι υπάρχουν κάποια πρότυπα που πρέπει να τηρούνται και στην περίπτωση του Πολωνικού Συμβουλίου αυτά τα, τα ελάχιστα πρότυπα, αυτές οι μήνυμου αρχές δεν τηρήθηκαν ε, για αυτό και δυστυχώς αποφασίσαμε να αποβάλουμε από το δίκτυό μας το Πολωνικό Δικαστικό Συμβούλιο και σας ε, ευχαριστώ. Πολύ σημαντική αυτή η αποβολή. Και όπως είπατε ήταν και ιδρυτικό μέλος το Πολωνικό Συμβούλιο και τα έχουμε ήδη αυτά συζητήσει και λεπτομερώ με τι αντιπροσωπείε σα. ευχαριστώ λοιπόν που τα εξηγήσατε ξανά και σήμερα λεπτομέρω για του συναδέλφου. Η αντιπροσωπεία μας στην Βαρσοβία ξεκίνησε με τον Άνταμ τον Βότμαρ, τον Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ήταν μια πάρα πολύ σημαντική συνάντηση. Οπότε χαίρομαι που ήρθε εδώ στην Ακρόαση και πραγματικά αναμένω να ακούσω αυτό το οποίο έχετε να μας πείτε. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου απευθύνατε να έρθω σε αυτήν την ακρόαση. Εκπροσωπώ τον συνηγόρο του πολίτη που έχει 30 χρόνια ιστορίας στο πολωνικό συνταγματικό σύστημα και βεβαίως στόχο μας είναι να βλέπουμε τι καταγγελίε και να προστατεύουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Πολωνία. Θεωρώ ότι ο ρόλος μας είναι να αντιδρούμε όταν το σύστημα προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων κινδυνεύει. Η εξέταση νομοθεσία από τα δικαστήρια αλλά και η λειτουργία των δικαστηρίων είναι πάρα πολύ κρίσιμη για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα ήθελα να τονίσω πω είμαι υπέρ ε, τη ε, μεταρρυθμίση τη πολωνική δικαιοσύνη, γιατί χρειάζεται μια μεταρρυθμίση για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των δικαστηρίων. Όμω ε, πρέπει να γίνει αυτή με σεβασμό στο κράτος δικαίου και δεν θα πρέπει να δικαιολογούνται αλλαγέ που επηρεάζουν την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και την διάκριση των εξουσιών. Γιατί σε τελική ανάλυση τα πραγματικά θύματα αυτών των αλλαγών είναι οι πολίτες μεταξύ των οποίων οι μειονότητες ε, και όσοι θέλουν μια ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Όσον αφορά το κράτος δικαίου. Ε, ενεργοποιούμε και στις περιπτώσεις των δικαστών οι οποίοι υφίστανται πιέσεις και κατά την απόψή μου το σημαντικότερο πρόβλημα και ο κίνδυνος στην Πολωνία είναι η έλλειψη ε, μιας ε, ανεξάρτητης δικαστικής εξέτασης των πραγμάτων. Είχαμε λοιπόν αυτά τα οποία ανέφερε ο καθηγητής ο κύριος Σόλτσεμ και τα οποία σχολιάζουν οι εκθέσεις της ε, Επιτροπής της Βενετίας που δείχνουν ότι οι δικαστές ε, δεν μπορούν ε, να δράσουν ανεξάρτητα ειδικά σε πολιτικοποιημένες υποθέσεις. Έχουμε λοιπόν κάποιους νόμους οι οποίοι συγκεντρώνουν την κρατική εξουσία και αφορούν την εισαγγελία, τις ε, αρμοδιότητες παρακολούθησης αλλά και νόμους περί μιμίες. Στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να αναφέρω δύο συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας. Η μία αφορά τις ε, διατάξεις ε, της εισαγγελίας και η άλλη αφορά τις αρμοδιότητες παρακολούθησης από την αστυνομία και τις μυστικές υπηρεσίες και πρέπει να πω ότι οι συστάσεις αυτές δεν εφαρμόστηκαν καθόλου Οπότε σε μεγάλο βαθμό αγνοήθηκαν παρά τις εκκλήσεις της δικές μου και της κοινωνίας των πολιτών. Θα ήθελα να πω ότι υπάρχει μια ενδιαφέρουσα κατάσταση με τα δημόσια μήμια. Έχουμε μια απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου από το 13 Δεκεμβρίου 2016 που βρήκε πως ο νέος κανονισμός περί δημοσίων ΜΜΕ που παρακάμπτει τις αρμοδιότητες του ΕΣΟΡΟΥ παραβιάζει το Σύνταγμα. Όμως η απόφαση αυτή του δικαστηρίου δεν εφαρμόστηκε. Ε, γιατί βεβαίως ε, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία εν ώψη και των ευρωεκλογών. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε κάτι το οποίο συνδέεται άμεσα με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Θεωρώ ότι ήταν σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει κάποια νομική δράση όσον αφορά ακριβώς το θέμα της παραβίασης της ανεξαρτησίας των δικαστηρίων. Κάτι το οποίο είχε μεγάλη σημασία για την ανεξαρτησία του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Γιατί ως αποτέλεσμα του προσωρινού μέτρου της, ε, του Οκτωβρίου του 2018 22 δίκαστες επανήλθαν στα καθήκοντά τους. Βεβαίως ε, υπάρχει το ζήτημα του εάν επαρκεί το κοινοτικό δίκαιο για να επανέλθουν οι δικαστές αυτές, αυτοί στα καθήκοντά τους. Σε συνδυασμό όμως με το πολωνικό σύνταγμα σίγουρα επαρκεί. Αλλά για λόγους αφήνειας θα πρέπει να υιοθετηθούν οι απαραίτητες νομοθετικές αλλαγές, οι οποίες όμως θα πρέπει να έχουν κάποιες πολύ απλές διατάξεις να λένε ότι είναι άκυρες οι νέε διατάξει περί συνταξιοδότησης και να επαναβεβαιώνουν ότι οι δικαστές αυτοί έχουν δικαίωμα να δικάζουν υποθέσεις. Θα ήθελα όμως να τονίσω ότι αυτό είναι ένα από τα πολλά προβλήματα με το κράτο δικαίου στην Πολωνία βεβαίω. Το θέμα του Ανωτάτου Δικαστηρίου είναι το πιο σημαντικό και συμβολικό. Α, το θέμα δεν είναι μόνο η ηλικία συνταξιοδότησης των δικαστών και η προστασία του Ανωτάτου Δικαστηρίου, γιατί βεβαίως σημασία έχει και ο σεβασμός των αξιών που μας προστατεύουν από τις αυθαιρεσίες της εξουσίας. Και εδώ πέρα θα ήθελα να αναφερθώ ακριβώς στο καστός του Συμβουλίου της Δικαιοσύνης. Ο κύριος Κιωστάρκ ανέφερε και επεκτάθηκε ακριβώ διάφορους νόμους που αφορούν το Εθνικό Συμβούλιο Δικαιοσύνης. Και ως αποτέλεσμα αυτού οι δικαστές μέλη, δηλαδή τα 15 από τα 20 μέλη, τώρα ορίζονται από τα 3 πέμπτα του Κοινοβουλίου και όχι από τους συναδέλφους τους. Και στις δημόσιες δηλώσεις μου στο Κοινοβούλιο εξέφρασα την επίσημη γνωμοδότηση ότι είναι αντισυνταγματική αυτή η μέθοδος ε, επιλογής. Επίσης αυτή ήταν η άποψη και πολλών λογίων ε, και δικαστών. Και εδώ πέρα θα ήθελα να αφαιρθώ ειδικά τον καθηγητή Άνταμ Τσέμπος, ε, ο οποίος ε, είναι και ένας Πολωνός ήρωας ε, και είχε ακριβώς θεμελιώσει το 1989 το σύστημα το δικαστικό και ήταν δική του η άποψη ότι θα πρέπει οι δικαστές να επιλέγονται από τους συναδέλφους του για να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ των εξουσιών. Αλλά Δυστυχώς η αλλαγή αυτή έγινε και τα νέα μέλη εξελέγησαν με τρόπο αδιαφανή και όλοι οι υποψήφοι μπορούσαν να υποβάλουν υποψηφιότητα με την σύσταση 25 συναδέλφων, αλλά μέχρι σήμερα δεν ξέρουμε ποιος στήριξε αυτούς τους υποψηφίους. Και βεβαίω, παρά τα μέτρα τα οποία έχει διατάξει το Ανώτο Διοικητικό Δικαστήριο υπάρχει μεγάλη δυσπιστία για τη λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Δικαιοσύνης και γι' αυτό ακριβώ ε, αποβλήθηκε από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο. Θεωρώ όμως ότι πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα στο καταστατικό του Εθνικού Συμβουλίου Δικαιοσύνης ε, γιατί έχει μεγάλο ρόλο στον ορισμό των δικαστών. Είναι ένα όργανο το οποίο αποτελεί μια δικλίδα ασφαλείας και πρέπει να είναι ανεξάρτητο. Θα ήθελα όμως να αναφέρω τις σοβαρές ανησυχίες που υπάρχουν για τα πειθαρχικά μέτρα κατά δικαστών. Σύμφωνα με τον ε, νέο κανονισμό δημιουργήθηκε ένα νέο σύστημα πειθαρχικού ελέγχου. Υπάρχει ο πειθαρχικός δικαστής ο οποίος ορίζεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης με σταθερή θητεία, ο οποίος μπορεί να δρά ατομικά αλλά και μέσω των βοηθών του που επίσης ορίζονται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Την εκτελεστική εξουσία δηλαδή στην ε, περίπτωση που έχουμε κάποια πειθαρχικά μέτρα, μετά έχουμε το εφετείο και κατόπιν ως ε, τρίτο βαθμό το ανώτο δικαστήριο. Και βεβαίως ε, δημιουργήθηκε το νέο αυτό πειθαρχικό τμήμα του ανωτάτου δικαστηρίου, το οποίο στελεχώθηκε με νέους δικαστές, οι οποίοι πληρώνται μάλιστα 40% περισσότερο από τους άλλους δικαστές του ανωτάτου δικαστηρίου και ω συνηγό του πολίτη παρακολουθώ κάθε πειθαρχική υπόθεση ει βάρο δικαστών που μπορεί να θεωρηθεί ότι ακριβώς επηρεάζει την δικαιοσύνη. Έχουμε λοιπόν αυτές τις ε, περιπτώσεις των 8 δικαστών. Θα ήθελα όμως ε, να σας δώσω μια γενική εικόνα. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις στην φάση των εξηγήσεων που είναι ε, πιθανό να πάνε στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, μόνο και μόνο επειδή έκαναν κάποιο προδικαστικό ερώτημα στο 10 σημαίνει ότι κινήθηκε εναντίον τους πειθαρχική διαδικασία. Τέσσερις άλλοι δικαστές ε, ελέγχονται πειθαρχικά γιατί σχολίασαν στα ΜΜΕ τις μεταρρυθμίσης της κυβέρνησης. Οι δικαστές ψημοσύνης και του Λέγια, Φρανσκόβιακ και ο Μάρκεβιτς, ο επικεφαλής της Ένωσης Δικαστών Γιουστίτσια. Με ενημέρωσε ο πειθαρχικός δικαστής ότι ζητήθηκε να καταθέσουν οι δικαστές αυτοί. Οπότε ε, πήγαν για ανάκριση και σε μία από αυτές τις ανακρίσεις ένας δικηγόρος που εκπροσωπούσε τους δικαστές, ο κύριος Γιάτσικ Τιπουά, αποκλείστηκε από την διαδικασία. Οπότε έχουμε μια νέα περίπτωση από αυτήν την κατάσταση. Επίσης υπάρχει και μια περίπτωση που αφορά ε, κατάσταση στην οποία ένας δικαστής αναφέρθηκε στην ε, τρέχουσα πολιτική κατάσταση και κάποιες επιδοτήσεις σε σχέση με ε, την σύζυγο ενό πολιτικού τη και αφορά τον δικαστή Σλάβο Μυρνιέτς. Μία άλλη περίπτωση αφορά τους δικαστές Φραντσκόβιακ και Κρούπα. Υπάρχουν λοιπόν διαδικασίες και αφορούν την χρήση της επίσημης ενδυμασίας τους σε μια προσωμείωση δίκης και αυτό θεωρήθηκε αιτία για πειθαρχικό έλεγχο. Θα ήθελα όμως να αναφέρω ότι υπάρχουν και πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις για τον Βάλτε Μαρζούρεκ, ε, ο οποίος ε, εργάζεται στο Περιφερειακό Δικαστήριο της Κρακοβίας. Ε, μετακινήθηκε παρά την θέλησή του από το εφετείο στο πρώτο δικείο και όπως σας είπα αυτό έγινε χωρίς να θέλει αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι ο ανώτερός του είναι ταυτόχρονα μέλος ε, του Εθνικού Συμβουλίου για την Δικαιοσύνη και υπάρχει ο κίνδυνος η υπόθεση αυτή να έχει πολιτική φύση. Ο Βάλτεκ Μαζούρεκ επίσης έχει ε, υποβάλει μήνυση κατά του Προέδρου του Δικαστηρίου της Κρακοβίας λέγοντας ότι υφίσταται παρενόχληση. Οπότε, πρώτα απ' όλα, οι διαδικασίες αυτές βρίσκονται στη φάση της διερεύνησης, αλλά το πολιτικό πλαίσιο του να ξεκινούν τέτοιες διαδικασίες κατά των δικαστών σημαίνει ότι οπωσδήποτε επηρεάζεται η συμπεριφορά του Σύμφωνα με μια δημοσκόπηση χιλίων δικαστών της Προσπολίτα τις εφημερίδες, ε, πάνω από 60% θεωρούν ότι αυτό θα επηρεάσει τη δουλειά του και 90% λένε ότι αυτή τη στιγμή απειλείται η ανεξαρτησία τη δικαιοσύνη. Δεύτερον, κανένα δικαστή δεν θα πρέπει να υφίσταται πειθαρχικό έλεγχο ε, για προδικαστικά ερωτήματα προς το 10. Τρίτον, υπάρχει το ερώτημα του εάν η ύπαρξη των ειδικών πειθαρχικών διαδικασιών με συμμετοχή της εκτελεστικής εξουσίας ε, είναι σύμφωνη με το άρθρο 19 της συνθήκης ε, και μία από τις πρώτες παραπομπές ε, προς το 10 ακριβώς αφορά αυτό το ζήτημα. Και τέλος το τέταρτο, η ύπαρξη του πειθαρχικού συμβουλίου του Ανωτάτου Δικαστηρίου δημιουργεί τον κίνδυνο πειθαρχικών κυρώσεων κατά δικαστών που είναι κατά των μεταρρυθμίσεων αυτών ή εκδίδουν αποφάσεις που δεν είναι αρεστές ε, προς ε, την πολιτική διοίκηση. Λοιπόν, πρέπει να λάβουμε υπόψη κάποια ζητήματα στην Πολωνία. Πρώτον, υπάρχουν περιορισμένες δυνατότητες άσκησης ε, δικαστικού ελέγχου της νομοθεσίας. Δεύτερον, θα έχουμε την εφαρμογή των συστάσεων της Επιτροπής της Βενετίας. Τρίτον, η εφαρμογή της απόφασης του Συνταγματικού Δικαστήριου για τα δημόσια ΜΜΕ, ειδικά εν ώψη και των ευρωεκλογών και την ανάγκη να υπάρχει ένας ανοιχτός και πλουραλιστικός διάλογος ε, στην προεκλογική εκστρατεία. Το επόμενο είναι το καταστατικό του Εθνικού Συμβουλίου Δικαιοσύνης και αξιολόγησή του και κατόπιν θα πρέπει να υπάρξει ένας έλεγχος των πειθαρχικών διαδικασιών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Μπότναρ. Θα δώσουμε τώρα τον λόγο στους ε, συναδέλφους για ερωτήσεις. Ξεκινάμε και πάλι με την σειρά με την οποία ζήτησαν τον λόγο οι συνάδελφοι. Ξεκινάμε τον κύριο Μπόνι. Δύο λεπτά, παρακαλώ. Μέχρι δύο λεπτά. Θα μιλήσω πλάνικα. Ευχαριστώ για τις διευκρινήσεις, ήταν σαφέστατες. Ευχαριστώ για την περιγραφή της κατάστασης. Ε, ερώτηση στον κύριο Πότνα. Πώς γίνεται όλες αυτές οι αλλαγές, μερικές δυσνόητες, πώς επηρεάζουν εν τέλει το σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην Πολωνία. Γιατί έχουμε ένα σωρό διαδηλώσεις πολλές φορές ε, απολύτως ε, ειρηνικές. Κι όμως ε, μαζεύεται η αστυνομία, τους μαζεύει, τους ανακρίνει. Έχουμε μια κατάσταση όπου οι ΜΚΟ βρίσκονται υποπίεση. Δηλαδή, περιορίζονται οι πόροι τους, δυσκολεύεται η έκφρασή τους. Και τούτο διότι, όπω είπε και ο πρόεδρο Ντούντα, προάγουν, λέει, την ομοφιλοφιλία στην Πολωνία. Η Πολωνία, εντάξει, είναι μια συντηρητική χώρα. Δεν μιλάμε εδώ τώρα όμω για ριζοσπαστικά κινήματα, για ακραία κινήματα, αλλά έχουμε και κάποιου νόμου. Πού πάνε αυτοί οι νόμοι μετά από όλε αυτέ τι αλλαγέ. Κύριο Γιουρέκ. Έω δύο λεπτά, υπενθυμίζω. Προνικά και εγώ. Πρόεδρε, ερώτηση είπα τον Υπουργό, τον κύριο Μπότνερ. Να ρωτήσω το εξή. Μάλλον μπορείτε να σχολιάσετε κάτι να πείτε όσον αφορά τον Πολωνό Επίτροπο, συνήγορο του πολίτη. Εδώ έχουμε μερικά εντάλματα σύλληψης κατά εγκληματιών τα οποία δεν εκτελούνται. Ενώ η δικαιοσύνη υποχρεούται να συνεργαστεί με τον εισαγγελέα βάση και τη συνθήκη για να προστατεύσει τους ε, Πολωνούς πολίτες. Και μπορεί. το λέω αυτό γιατί δεν γνωρίζουν όλη την πολιτική νομοθεσία. Γιατί ε, στη χώρα μας το Σύνταγμα αποσκοπεί και στην προστασία της ζωής των πολιτών. Το έχει πει αυτό και το Συστηματικό Δικαστήριο. Και αυτά τα λέει και η Ευρωπαϊκή Ένωση με διάφορε δηλώσει που έχουν γίνει κατά επανάληψη κλπ. Λοιπόν, δεν πρέπει να γίνει σεβαστή και η πολωνική νομοθεσία και στην Ευρώπη. Επαναλαμβάνω, αυτό είναι και το καθήκον της πολωνικής δικαιοσύνης. Και ρωτώ τον Κλοντ και του ζητώ να πει κάτι. Ε, όχι τώρα αναγκαστικά, δεν θέλω μια απάντηση τώρα, αλλά ε, για σκέψτε το λίγο. Δεν νομίζω ότι τέτοιες δηλώσεις πρέπει να γίνονται εδώ. Και βάσει ε, του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορεί να διαφωνούμε όσον αφορά την οικογένεια, και τα οικογενειακά ζητήματα. Ε, και δεν σημαίνει ότι όταν κάποιο διαφωνεί είναι ρατσιστή. Οπότε παρακαλώ, πείτε δύο λόγια. Ελπίζω να μην έχουμε άλλε τέτοιε ε, ακραίε αντιδράσει εδώ. Ευχαριστώ. Um, uh, να πω Μετά την παρέμβαση αυτή θα παρέχω στην Προεδρία, στον κύριο Κιλάρο. Παρακαλώ, αφού μιλήσετε. Αλλά πρώτα κύριε Σπινελή, δύο λεπτά, υπενθυμίζω. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε την Επιτροπή της ε, Βενετίας αλλά και το Δίκτυο Δικαστικών Συμβουλίων. Επίσης, ιδιαίτερω να ευχαριστήσουμε τον Πολωνό την Μπόντναρ, ο, ο οποίος ε, δέχεται πειρά όλη αυτή την περίοδο. Έχω διαβάσει πολλές από τις ε, γνωμοδοτήσεις σα και δεν διέκρινα πολιτικοποίηση για την οποία κατηγορείστε. Πάντως, υπάρχει πολιτικοποίηση σε ό,τι προβάλλεται ως ε, αιτία ελαττήριο αυτών των μεταρρυθμίσεων. προβάλλεται ως ε, πρόφαση η αποκομμουνιστικοποίηση της διοίκησης. Ε, αυτό δεν είναι φορτισμένο ιδεολογικά. Δεύτερον, Αυτές οι μεταρρυθμίσεις στην δικαιοσύνη αναβαθμίζουν τις αρμοδιότητες της κυβέρνησης. Και ε, τελικά έχει συγχωνευτεί η εισαγγελία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Πάντως αυτό είναι γενικότερο φαινόμενο, δεν γίνονται αυτά μόνο στην Πολωνία. Τον Ιανουάριο φέτος ο πρόεδρος Μακρόν μετά πολλές δεκαετίες πολεμικής για την αμφισβήτηση ανεξαρτησίας της Γαλλικής Αγγελίας είπε ότι οι σχέσεις μεταξύ τελικής εξουσίας και εισαγγελίας θα πρέπει να είναι ισχυρές και ότι ο ίδιος είναι κατά της ανεξαρτησίας που οι περισσότεροι από τους δημοκράτες δικαστές είχαν ζητήσει. Αυτά. Θα πρέπει να μας πει τη γνώμη για τις άλλες χώρες, γιατί νομίζω ότι αυτό το φαινόμενο της ενίσχυσης κυβέρνησης βάρος της δικαιοσύνης γίνεται και αλλού. Εμείς ευχαριστούμε κύριε Αφινέλη, λέει ο πρόεδρος και τώρα κύριε Γκόμες έχει το λόγο. Ε, ευχαριστούμε όλους τους ε, προσκεκλημένους μας τα είπαν εξαντλητικά, ενημερωτικά και έτσι μπορούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Ε, βέβαια τώρα ανησυχώ ακόμα περισσότερο. Τώρα που σας άκουσα. Γιατί. Διότι. Δεν υπάρχει πια ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Δεν λειτουργούν πια ασφαλιστικές ε, δικλείδες. Πολύ εύγλωτα το μας τα εξηγήσατε. Και γιατί ανησυχείτε. Αν μου δίνετε νωρίτερα το λόγο, θα έλεγα αυτό που θα σας πω τώρα, κυρίως για να απαντήσω στον κύριο Γιούρεκ. Όχι! Δεν πρόκειται περί επίθεσης κατά του πολιτικού και της Πολωνίας. Το αντίθετο. Επειδή εκτιμούμε, σεβόμαστε τους Πολωνούς και την ε, Πολωνία. Ξέρουμε ότι είναι πολύ ζωντανή η κοινωνία σας. Ψηλό επίπεδο και γι' αυτό θέλουμε να σας διέπουν τα καλύτερα δυνατά πρότυπα. Ε, αυτά δεν είναι όμως ε, ε, πρότυπα αυτά που γκρεμίζουν το κράτος δικαίου. Πάρα πολύ κακό για την εικόνα της χώρας, της δικαιοσύνης που δεν απονέμεται ούτε οι ανθρώπινα δικαιώματα τηρούνται και βέβαια είναι πάρα πολύ κακό και για την φήμη των επιχειρήσεων. Γιατί πάρα πολλοί που κάνουν δουλειά στην Πολωνία το κάνουν επί τη βάση του ότι λειτουργεί το κράτος δικαίου. Ε, με τέτοια πολιτικοποίηση περιμένουν το χειρότερο. Ακατανόητο μου φαίνεται που η κυβέρνηση δεν κάθε στο τραπέζι να τα συζητήσει. Δεν το κάνει ούτε με εμάς ούτε με την Κομισιόν. Απαράδεκτο. Όση φορά Ακούω πολλές ε, δικαιολογίες, ο κίνδυνος του να έχουμε διάχυση των ομοφιλοφιλικών ε, αξιών. Μα τι πράγματα είναι αυτό. Μα τι είναι αυτά, κάνουμε σαν τον Πούτιν φανατισμός, μίσος, αυτά εξαπλώνονται. Τι έγινε με χριστιανικές αξίες της Πολωνίας. Τι να σου πω, έχουμε μείνει το στόμα ανοιχτό. Thank you, Mrs. Gomez. Ευχαριστώ κυρία Γκόμες. Κύριο Σκάρσκι. Ευχαριστώ πρόεδρε. Παρακολουθώ τη συζήτηση και η εντύπωση μου είναι ότι τα πράγματα δεν είναι και πολύ ισορροπημένα. Ο κύριος Μπόναρ τα είπε πιο σωστά, πιο ισορροπημένα από όλους. Βέβαια τις απόψεις του είπε, αλλά ήταν πιο μητριοπαθής. γενικά. Σε κάθε χώρα που υπάρχει διαίρεση των εξουσιών και διάκριση των εξουσιών, αλλά τι γίνεται όταν κατεβαίνουν σε διαδηλώσεις πολιτικού περιεχομένου οι δικαστές, τι γίνεται όταν ε, εκφράζουν πολιτικές απόψεις, τι κάνουμε όταν βγαίνουν σε τηλεοπτικές εκπομπές και τσακώνονται για τα πολιτικά με πολιτικούς. Α, ο δικαστής Ζούρεκ καλείται σε εκπομπές και τσακώνεται με πολιτικούς και άλλους. Τι κάνουμε επομένω όταν οι δικαστές πηγαίνουν σε πολιτικές συγκεντρώσεις της αντιπολίτευσης και όταν ε, κάνουν ομιλίες για το πώς θα έπρεπε γενικώ να οργανωθεί η χώρα και το κράτος. αυτό υπονομεύει την διάκριση των εξουσιών. Ο δικαστής, θα πρέπει να εκφράζεται μέσω των δικαστικών αποφάσεων. Τότε είναι δικαστής. Δεν θα πρέπει να ασκεί πολιτική δραστηριότητα. Καλά, σε κάποιες χώρες επιτρέπεται να είναι με ελικόματος όπως στην Γερμανία. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι λάθος και θα πρέπει να αλλάξει. Θα πρέπει να είναι απολύτικοι οι δικαστές στην Πολωνία. Απαγορεύεται ο δικαστής να είναι μέλος κόμματος. Απαγορεύεται να σκούν πολιτική δραστηριότητα. Ούτε μπορεί να είναι συνδικαλισμένοι. έχουν αυτό τον φορέα τους, ούτω ώστε να προστατεύονται τα του επαγγέλματος τους. Άρα θα πρέπει η συζήτηση να γίνει ισορροπημένα. Ελέγχθη ότι υπάρχει ταύτιση Υπουργή Δικαιοσύνη και Εισαγγελία με αυτό ισχύει σε πολλέ χώρε. Και ισχύει και στην ε, Πολωνία του 2015. Παλιότερα υπήρχε διάκριση. Ο επόμενο. Πρόεδρε. Ναι, το ξέρετε, είναι κουραστικέ αυτέ οι συζητήσει. Είναι διάλογο κοφών γιατί έχουν ακουστεί πολλά επιχειρήματα από ειδικού, ανεξάρτητους και η αντίδραση από τους Πολωνούς εθνικιστές είναι πάντα ίδια. Πρώτα λένε είναι άδικο, δεν μας σέβονται, δεν μας ακούνε» και μετά αρχίζουν να λένε άλλες χώρες «Α, ναι και άλλες χώρες κάνουν το ίδιο» γιατί δεν προβάλλεται κάποιο αντιεπιχείρημα ουσιαστικό. Αντί να κάθεστε εδώ πέρα και να παριστάνετε το θύμα. Δεν είστε εσείς το θύμα. Δεν είστε θύμα. Εσείς υπονομεύετε την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και θα επαναλάβω αυτό το οποίο πριν δεν έχει σχέση με το δικαίωμά σας να έχετε άποψη κύριε Γιούρο. Έχετε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που προβλέπει την υπονόμευση όχι μόνο της δικαιοσύνης αλλά τα δικαιώματα των γυναικών, ελευθερία των ΜΜΕ, μπελοάτκι, ε, πλουραλισμό και όλα αυτά. Αυτό επισημαίνω. Οπότε μην παριστάνετε το θύμα, δεν είστε το θύμα το ερώτημά μου τώρα προς το πάνελ. Ε, πρώτη ερώτηση. Έχουν υπάρξει κάποια ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης που έχουν εκδώσει Πολωνοί δικαστές και νομίζω ένας Ιρλανδός, ένας Ολλανδός και ένας Γερμανός δικαστής, αρκετοί δικαστές, αρνήθηκαν να τα εκτελέσουν. Νομίζω ότι ο Ιρλανδός ο δικαστής εντωμεταξύ τελικά το εκτέλεσε, δεν είμαι σίγουρη. γνωρίζετε εσείς άλλες τέτοιες ε, περιπτώσεις. Ε, ε, θεωρείτε ότι θα γίνουν τα πράγματα χειρότερα, πώς το βλέπετε. Και η δεύτερη ερώτηση είναι. Οι εθνικιστές λένε μα αυτό το οποίο κάνουμε εμείς δεν είναι τίποτα σπουδαίο για το κάνουν και σε άλλες χώρες. Να δείτε τη Γερμανία, τι φοβερό, τι τρομερό, πολιτικοί δικαστές. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν στοιχεία στο πολωνικό σύστημα που υπάρχουν και σε άλλες χώρες. Αλλά με τελείω, σε τελείως διαφορετικό πλαίσιο. πολύ ισχυρότερες δικλείδες ασφαλείας. δεν ξέρω λοιπόν αν μπορείτε να μας πείτε κάτι για να αντικρούσετε αυτά τα πλουστευτικά επιχειρήματα των συνάδελφων. Πιτέλα πριν επανέλθουμε στο πάνελ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να απαντήσω στον κύριο Κάρσκι που λέει ότι οι δικαστές δεν ε, χρηματοδοτούν ενώσεις ε, που αντιμάχονται. Δεν ίδρυσαν ενώσεις δικαστών για να πολεμήσουν την κυβέρνηση. Αυτές οι ενώσεις υπήρχαν. Ενώσεις οι οποίες εκπροσωπούσαν τους ε, δικαστές ε, εδώ και καιρό. Δεν είναι κάποια συνωμοσία λοιπόν. Αλλά γιατί είναι παρόντες οι δικαστές στην τηλεόραση. Να υπενθυμίσω στον κύριο Κάρσκι ότι ο νυν πρόεδρος του συνταγματικού δικαστηρίου είναι πολύ παρόν στα δικαστήρια και κάνει και δηλώσεις που μπορούν να θεωρηθούν πολιτικές. Το συνταγματικό δικαστήριο υπονομεύθηκε όπως και το ανώτατο δικαστήριο και όλα έχουν αλλάξει γενικώ τα αστικά δικαστήρια Επίσης ε, έχουν ξεθεμελιωθεί και ε, μέλη της οικογένειας ε, των πολιτικών τοποθετούνται σε διάφορες δέκο και η χρηματοδότηση των ΜΚΟ από το κράτος έχει αλλάξει και ακούμε συνεχώς για τα προβλήματα των δημοσίων ΜΜΕ και υπάρχει το σύνθημα της ε, επαναπολωνοποίησης ε, των ε, ΜΜΕ που είναι υποξένη ιδιοκτησία και δεν χρειάζεται να σας πω τι έγινε με την δημόσια τηλεόραση. Το αντιλαμβάνεστε. Η ΜΜΕ, τα, οι ε, βουλευτέ μα συγχωρείτε τη αντιπολίτευση περιγράφουν σαν ΜΜΕ με πολύ ακραίο τρόπο. Θα ήθελα λοιπόν να προσθέσω μόνο κάτι ακόμα και θα ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Μπόντναρ να το σχολιάσει γιατί τίποτα δεν ακούσαμε ακριβώς για το θέμα αυτό με τους Πολωνούς Ευρωβουλευτές όταν ο πρόεδρος του κόμματος αποφάσισε ότι η μισθή των βουλευτών θα κοβόταν στο μισό. Και ο πρόεδρος του Πολωνικού Κοινοβουλίου όταν κάτι δεν του αρέσει μπορεί να κόψει το μισθό του οποιοδήποτε βουλευτή στο μισό και να υπάρχει δικαίωμα προσφυγής. Οπότε κύριε Γιούρεκ, εάν λέτε ότι αυτά που συμβαίνουν εδώ πέρα είναι λάθος, με ποιο κοινοβούλιο το συγκρίνετε, γιατί ο κύριος Κόρβιν Μικέ προσέφυγε σε δικαστήριο και ε, του έδωσαν πίσω τα λεφτά του. Και όλοι ξέρουμε το τι συμβαίνει στο Πολωνικό Κοινοβούλιο. Ε, δεν θα πρέπει λοιπόν να προσβάλλετε το τι συμβαίνει εδώ. Ε, βεβαίως αντιλαμβανόμαστε τα ευαίσθητα ζητήματα. Θα θέλαμε όμως οι Πολωνοί συνάδελφοι να μην ε, κάνουν ε, οριζόντιες ε, τοποθετήσεις και ανταλλαγές απόψεων. Λοιπόν, Θα σας δώσω 30 δευτερόλεπτα για να απαντήσετε και μετά θα επανέλθουμε στους ομιλητές ε, του πάνελ. Παρακαλώ. Κύριε Κάρσκι, σας ευχαριστώ. Η συνάδελφος ανέφερε την δήλωσή μου. Ε, εγώ είμαι εδώ από την αρχή. Α, δεν σας είχα προσέξει. Τέλο πάντων, δεν το έκανα επίτηδε. Ήθελα να πω κάτι για τις πολιτικές δραστηριότητες κάποιων Πολωνών δικαστών. Και ήθελα να αναφερθώ στους ε, δικαστές ε, που βγάζουν ε, αποφάσεις χωρίς να αναφερθώ στις μηντιακές δραστηριότητες εκπροσώπων ή προέδρων δικαστηρίων ή του πρώτου πρόεδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Γιατί αυτοί έχουν διοικητικές, διοικητικά καθήκοντα. Ένας κανονικός δικαστής λοιπόν, ο οποίος υποτίθεται ότι είναι ανεξάρτητος. Πηγαίνει σε διαδηλώσεις ε, και εκφράζει πολιτικές απόψεις. Ε, δεν είναι πλέον αμερόληπτος και δεν μπορεί να θεωρείται αμερόληπτος. Ε, ας μην ξεκινήσει ξανά η συζήτηση. Λοιπόν, επανερχόμαστε στο πάνελ. Κάποιοι βουλευτές πρέπει να φύγουν μέχρι τις 5, ο κ. Γιούρεκ δηλαδή. Δεδομένου του ότι ερώτησε συγκεκριμένα και ζήτησε κάτι από τον κύριο Μπόντνερ. Προτείνω να ξεκινήσουμε με την αντίστροφη σειρά. Ακούσουμε πρώτα τον κύριο Μπόντνερ και μετά τους υπόλοιπους. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις. Να απαντήσω πρώτα στον κύριο Γιούρεκ. Πρώτα απ' όλα υπάρχει απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τον κύριο Τσέ. Αφορούσε την έκδοση από την Ελλανδία στην Πολωνία. Μια κλασική υπόθεση του τι πρέπει να κάνει ένα δικαστήριο προκειμένου. Οι δικαστές στην Ισπανία, στην Ολλανδία, άρχισαν να θέτουν κάποια ερωτήματα προσπαθώντας να πούν ότι δεν μπορείς να εκτελέσεις ένα ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης αν δεν πληρούνται κάποιες συνθήκες. Χθε ο δικαστής Ντόναλες στην Ιλλανδία έλαβε απόφαση ε, ο οποίος αφού έλεγξε την κατάσταση, έκανε τη δική του διάγνωση, οι δικαστής εξετάζοντας και το κατά πόσον τηρείται το τεκμήριο της αθόρυτας, αποφάσισε ότι μπορεί να παραδοθεί ο άλλο κρατούμενος στην Πολωνία. Ο δικαστής οφείλει να εξετάσει ποια είναι η κατάσταση στη χώρα προορισμού ούτως ε, Πίν. Αυτό είναι υποχρεωτικό. Τώρα για την προστασία της ζωής βάσει της πολιτική νομοθεσίας. Η πολιτική νομοθεσία εξασφαλίζει μια ισορροπία θα έλεγα μεταξύ αφενός της προστασίας της ζωής και αφετέρου της προστασίας διαφορών αξιών στην κοινωνία. Στην Πολωνία έχουμε τρεις δυνατότητες τερματισμού μια εγκυμοσύνης. Εγώ ως σύνολος του πολίτη πρέπει να Έξακριβώ, κατά πόσον τηρείται ο νόμος σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Όταν μια γυναίκα βρίσκεται σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν πληρούνται δηλαδή οι τρεις αυτές προϋποθέσεις για να διακοπεί η κοίηση, ώστε μια γυναίκα να έχει πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίε. Να μην υψέλθω τώρα σε λεπτομέρειες, Πάντω ε, δεν είναι ο ρόλος μου σε καμία περίπτωση να κρίνω κατά πόσον ο νόμος πρέπει να φιλελευθερωποιηθεί, να προχωρήσει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Τώρα, τι γίνεται με την δικαιοσύνη εν γέννη και ποιε είναι οι επιπτώσει επί των δικαιωμάτων. Είναι βέβαιο ότι η σημερινή κατάσταση ναι, επηρεάζει δικαιώματα και ελευθερίες. Υπάρχει μια συναισθηματική πτυχή προκειμένου ε, κάποιοι δικαστές πιέζονται και είναι αρκετές οι περιπτώσει που δεν είναι σαφές αν μια απόφαση έχει ληφθεί σύμφωνα με το Σύνταγμα, τους νόμους ή υπό πολιτικές ε, πιέσεις τις οποίες δέχτηκαν οι δικαστές ή αν ο δικαστής φοβάται κάποια πειθαρχική δίωξη. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν δεν μπορεί κανείς να είναι 100% βέβαιος ότι τηρήθηκαν όλα 100%. Πάντως, στη διάρκεια των χρόνων ε, θα μπορούσε να πει κανεί ότι η κατάσταση μάλλον θα επιδεινωθεί. Μία από τις μεταρρυθμίσεις πάντως ήταν η θέσπιση, η δημιουργία μάλλον αυτού του νέου σώματος ε, αναθεώρησης όλων των αποφάσεων των τελευταίων 20 ετών. Εκεί όντως υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, δηλαδή να επανεξεταστούν υποθέσεις που αφορούν ευάλωτε μειονότητες. Ο Γενικός Εισαγγελέας θα μπορούσε λοιπόν να τροποποιήσει ουσιαστικά την ομολογία επί συγκεκριμένων ζητημάτων που έχουν και μια ιδεολογική φόρτιση. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Όμως, η ιδιαίτερη αυτή κατάσταση, οφείλω να πω, δημιουργεί και μια ατμόσφαιρα του ΣΥΠΗΝ. Οι δικαστές μάλλον θα προσέχουν λίγο πιο πολύ το Σύνταγμα. Πιστεύω ότι έτσι θα έχουμε ενδεχομένω καλύτερε αποφάσει και για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Α πούμε, σύλληψη ε, προσώπων μετά από διαδηλώσει κλπ. Εδώ πιστεύω ότι έχουν μια ευκαιρία δικαστέ να αποδείξουν ότι είναι ανεξάρτητοι. Για αυτό που είπε ο κύριο Κανσκή όσον αφορά τη συμμετοχή σε διαδηλώσει. Να πω απλώ ότι κατά τη γνώμη μου είναι πρότυπο δικαιωμάτων του ανθρώπου το θέμα αυτό. Όπως όλοι οι πολίτες μπορούν να λαμβάνουν μέρος σε διαδηλώσεις, έτσι μπορούν και οι δικαστές. Και αν εσείς είστε με στα μεταδιεθνούς δικαίου, μπορώ να σας βεβαιώσω και εγώ για αυτό που μόλις είπα. Είναι θέμα κράτους δικαίου. Είναι απολύτως βέβαιο ότι οι δικαστές έχουν το δικαίωμα να διαδηλώνουν. Ο κύριος Σέμπος είναι 88 ετών, γνωρίζει το θέμα, είναι συνταξιούχος δικαστής και είναι ο δικαστής ο οποίος κατέβηκε σε διαδήλωση στην ηλικία αυτή. Νομίζω ότι πρόκειται μια απολύτως ηθική δεντολογική στάση. Και το τελευταίο και επιτέρα. Όσον αφορά το ρόλο της Βουλής. Στην Πολωνία το Κοινοβούλιο περιθωριοποιείται. Μειώνει το χρόνο αγόρευσης, θεσπίζονται διάφορα μέτρα, ε, με τα οποία τιμωρούνται επί της ουσίας οι βουλευτές. Έχουμε μια ενδιαφέρουσα απόφαση, η οποία πήγε ε, από τον κύριο Στέρμπα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η υπόθεση παρόμοια με την Καρατσόνη και άλλη κατά Ουγγαρίας. Στην περίπτωση που ένας βουλευτής τιμωρείται για τη δράση του στο Κοινοβούλιο, ε, στην Πολωνία υπάρχει δυνατότητα προσφυγής κατά του βουλευτή. Ε, ελπίζουμε όμω ότι η προσφυγή του βουλευτή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα έχει ευτυχή κατάληξη. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρο. Ο χρόνος δυστυχώ πιέζει τους πάντες και εσά για να περάσουμε στο επόμενο πάνελ, κύριε Στέρκ. Πέντε λεπτά. ξεχάσετε και στο χρόνο. Εγώ έχω δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη για την συμμετοχή των δικαστών στην πολιτική. Σύμφωνο με τον ε, κύριο Μπότνερ, ο κανόνας είναι απλό. Αυτό Περισμός. Όταν όμω κινδυνεύουν οι αξίε, τότε ένα δικαστή πρέπει να λάβει θέση. Και αυτό όχι μόνο στην Αμερικανική νομολογία, αλλά και στην Ευρωπαϊκή νομολογία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών επίση εξέδωσε γνώμη επί του συγκεκριμένου θέματος. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το θέμα δικαστές και πολιτική. Δεύτερον, για τα λεγόμενα στοιχεία για τα οποία έχει λάβει μέτρα η πολιτική κυβέρνηση για τη σύμπηξη του ρόλου του Γενικού Εισαγγελέα με το ρόλο του Υπουργού Δικαιοσύνη. Σε μερικέ χώρε συμβαίνει αυτό. Ε, Όπω επίση και τον ορισμό τη ηγεσία τη δικαιοσύνη. Ναι, ό,τι και να συζητήσουμε, ναι, υπάρχει κάτι παρόμοιο σε κάποια άλλη χώρα. Αυτό είναι αληθέ. Όμω, πρέπει να δει κανεί τη μεταρρυθμίση αυτή στο σύνολό τη. Τι μεταρρυθμίσει αυτέ, το σύνολο του, η οποία τελικά, οι οποίες μάλλον τελικά κατατείνουν σε έλλειψη δικλείδων ασφαλείας στο πολίτευμα. Και αυτό λέει και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο. Ότι στην Πολωνία έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα δεν υπάρχουν πλέον ασφαλιστικές δικλείδες στο πολίτευμα όσον αφορά τις εξουσίες και τη διάκρισή τους. Ευχαριστώ. Καθηγητά Σόλτσεν, κύριε Πρόεδρε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Να συνεχίσω το θέμα εκεί που το άφησε ο κύριος Στέρκ. Οι συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας ακόμα και στα πιο δύσκολα θέματα ακούγονται, γίνονται σεβαστές. Και γιατί αυτό. Διότι οι ομάδες των ειδικών που συγκροτούνται από την Επιτροπή ε, έρχονται από μια πολυσυλλεκτική ε, νομική κουλτούρα. Άλλοι καθηγητές, άλλοι δικαστές κλπ. Άρα πρόκειται για κάποιο είδου ποικιλία που γνωμοδοτεί. Ποικιλία των ούτε αποφαίνονται στενά για τα νομικά. Επομένως, αυτά τα προβλήματα είναι δύσκολα. Αλλά το πιο δύσκολο θέμα είναι το ζήτημα της εισαγγελίας γιατί εκεί υπάρχουν πολύ πιο μεγάλες αποκλήσεις στην Ευρώπη από το θέμα της ανεξαρτησίας των δικαστών. Τα προβλήματα μας απασχολούν είναι τεράστια. Να αυτή η ιδέα που εγκαταλείφθηκε ότι δηλαδή το συνταγματικό δικαστήριο δεν μπορεί να ακυρώσει έναν νόμο παρά μόνο αν έχει την ε, πλουσία των δύο τρίτων. Δεν ισχύει αυτό που θέλω. Και επίση το τελευταίο που θέλω να σας πω ως απάντηση είναι ότι σε αρκετές περιπτώσεις Μα είναι πολύ αξιόλογοι οι Πολωνοί δικαστές. Ξέρουν τι ισχύει στο εξωτερικό και μπορούν να συγκρίνουν να πούν ότι αυτό ξεχάστηκε, αυτό παραμελήθηκε. Να επομένω γιατί αξίζουν οι συστάσεις της υπηρεσίας της ε, Βενετίας. Γιατί συγκεντρώνει όλα αυτά τα διαφορετικά στοιχεία. Ξέρουν τους νόμους ε, για τα δικαστήρια, για την εισαγγελία κλπ. Όλους, όλους. Το έχει πει ο Μοντεσκέ. Ότι ε, ε, αναγκαστικά το μόνο πράγμα που φρενάρει την ε, εξουσία είναι η εξουσία. Επομένω και όλα αυτά τα οποία είναι στην Πολωνία, τι λέει η Επιτροπή τη Βενετία, λέει όχι. Σα ευχαριστώ όλου λέει ο κύριο Αγγιλάρ. Διακόπτουμε μέχρι να λάβουν θέσεις οι επόμενοι προσκεκλημένοι του επόμενου πανεπιστημίου. Alors, on va commencer dans le prochain panel. C'est le panel Academia Civil Society. We kindly invite our new speakers and guests to take their floor in the panel. Παρακαλώ. Λάβετε θέσεις στο πάνελ. Now, Όπως προβλέπετε ούτως ή άλλως, περνάμε στο τρίτο τη συνάντηση με εκπροσώπου του πανεπιστημιακού χώρου και τη Κοινή των πολιτών. Έχουμε τον καθηγητή Πέσο, καθηγητή Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Μίλσεξ του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, τον Ζήχ. Ζιχ, καθηγητή στην έδρα Θεωρία και Φιλοσοφία του δικαίου, στη νομική σχολή και διοίκησης στο Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας, τον κύριο Στέφαν Βυσίνσκι, τον κύριο Μάικλ Μαυρικίβιτς, δικηγόρο, όχι, δεν το, δεν το πρόφερα σωστά. Ε. Το έκανα τελείως λάθος, ε. συγγνώμη. Ε, δικηγόρο, Φολεσάντι, του κινήματος Ελεύθερα Δικαστήρια. Και έχουμε και την κυρία Μαλκοσάτα Σουλέκα, στο Ίδρυμα του Ελσίνκη για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Είμαστε εδώ, όπως γνωρίζετε, με την ευκαιρία, με, με αφορμή την επίσκεψη του κλιμακίου της Λίμπε στην Πολωνία. Έχουμε λοιπόν τον κύριο Πες, τον οποίο συνέντησε το κλιμάκι, τον κύριο Σίχ, τον κύριο βρικέβιτς. που αποτελεί γνώστη του τομέα. Λοιπόν, 8 λεπτά θα δώσω στον κάθε μιλητή. 8 λεπτά και μετά θα συνεχίσουμε και θα κλείσουμε με ερωτήσεις και απαντήσεις. Ο καθηγητής, ο κ. Σπέκ. Παρακαλώ, κ. καθηγητά. Να περάσω αμέσως στο θέμα, γιατί μου είχαν πει 10 λεπτά, θα τα κάνω 8. Αυτό παρακαλώ ναι. για όλους μας και για τους διερμηνείς και για όλους. Παίρνω στο θέμα χθε. Ήταν η εκπνοή της προθεσμίας για τις πολωνικές αρχές να συμμορφωθούν με την ενδιάμεση απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου όσον αφορά την πολωνική νομοθεσία για το ανώτατο δικαστήριο. Μάθαμε σήμερα με ενδιαφέρον ότι η πολωνική κυβέρνηση περιμένει την τελευταία μέρα να καταθέσει σχέδιο δράση αντί να μα πει συγκεκριμένα τι θα κάνει, ότι δηλαδή έκαναν αυτά που έπρεπε να κάνουν. Φαίνεται ότι προσπαθεί για άλλη μια φορά να κερδίσει χρόνο η πολωνική κυβέρνηση, κολλησιεργώντας αντί να συμμορφωθεί με τις απαιτήσει του κράτους δικαίου. Ο Πολωνός Πρόεδρος, αν είναι σωστές οι πληροφορίες μου, αντί να δηλώσει πώς η χώρα θα συμμορφωθεί αμέσως, μας λέει ότι το δικαστήριο υπερέβαλε αυτόν κλπ. Η αγνία του νόμου και περιφρόνηση στο δικαστήριο που αντιμετωπίζουμε στην Πολωνία είναι άνευ προηγουμένου. Επαναλαμβάνονται λοιπόν εν και αυτή τη απόφαση τα ίδια. Το δικαστήριο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, βλέπει με έκπληξη δυστυχώς την εκτελεστική εξουσία να αρνείται απλούστατα να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου όσον αφορά τον ορισμό των δικαστών στο ανώτερο δικαστήριο. Δυστυχώς, όπως είπα, αυτά τα έχουμε ξαναδεί και οι περισσότεροι ξεχνούν αυτήν την πτυχή του προβλήματος. Πρόκειται για την ίδια αρχή, την ίδια εκτελεστική εξουσία, η οποία και στο παρελθόν προτίμησε να αγνοήσει το Συνταγματικό Δικαστήριο και να μη συμμορφωθεί πριν αλλάξει η σύνθεση του Συνταγματικού Δικαστηρίου στο τέλος του 2016. Αυτό, κατά την γνώμη μου, είναι η σκληρή πραγματικότητα. Έχει πει και η Κομισιόν σε μια παλαιότερη συστασή τη. Και αυτή τη στιγμή είμαστε μάρτυρες μιας κατάστασης άνευ προηγουμένου. Έχουμε λοιπόν μια χώρα η οποία από το Δεκέμβριο του 2016 δεν έχει μηχανισμό ελέγχου της συνταγματικότητα της νομοθεσίας. Αυτό σημαίνει ότι η νομοθετική εξουσία και η εκτελεστική κάνουν ό,τι θέλουν, ό,τι τους βολεύει, ανεξαρτήτως του συντάγματο της Πολωνία. Αυτό, κατά την άποψή μου, είναι άνευ προηγουμένου. Και δικαιολογεί 100% την ενεργοποίηση του άρθρου 7 παράγραφος 1 τον Ιανουάριο του 2017. Κατά τη γνώμη μου η Επιτροπή θα έπρεπε να το έχει κάνει αυτό νωρίτερα γιατί τον Ιούλιο του 2017 διορθώνω ήταν κάτι παραπάνω από προφανές ότι υπήρχαν νομοθετήματα τα οποία δεν συνάδουν με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Από εκεί πέρα τα υπόλοιπα ήταν αναμενόμενα δηλαδή εγώ ως καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου και ως ειδικός περί τα νομικά επί πολλά χρόνια ε, θα ισχυριστώ εδώ ότι αυτά τα οποία είδαμε και πιστεύω και φοβούμε θα δούμε αποτελούν κατά συρροήν παράβαση του ευρωπαϊκού δικαίου. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε σήμερα. Σχεδόν τρία χρόνια μετά από την ε, ενεργοποίηση του άρθρου 7 Έχουμε τέσσερις συστάσεις. Μία φορά το 1 Αιτιολογημένη ε, σύσταση. Αν με ρωτήσετε, βελτιώθηκε η κατάσταση. Η απλή μου γρήγορη επάνηση είναι όχι. Μάλιστα θα έλεγα ότι επιδεινώθηκε η κατάσταση και έγινε χειρότερη από ποτέ. Η ενεργοποίηση του άρθρου 7 πρέπει να συνεχιστεί. Έχουμε πολλαπλά θέματα τα οποία παραμένουν ανεπίλητα. Δεν θα τα περιγράψω τώρα ένα προς ένα, ούτε μία προς μία τις συστάσεις, τις οποίες κατάφορα αγνοεί η πολωνική κυβέρνηση. Είναι πολλές αυτές οι συστάσεις, μεταξύ αυτών ίσως πιο σημαντική είναι αυτή που ζητάει από τις πολωνικές αρχές να συμμορφωθούν με τη σύσταση της Κομισιόν να αποκαταστήσουν την αξιοπιστία και την ανεξαρτησία του Ανώτατου Δικαστηρίου ως εγγυητή του πολιτικού συντάγματο. Δεν υπάρχει κρατό δικαίου σε ένα σύστημα όπου το σύνταγμα μπορεί να το παραβέζει ο καθένα όποτε θέλει και μάλιστα η εκτελεστική και η νομοθετική εξουσία. Αυτή είναι η διάγνωσή μου της κατάστασης στην οποία συμμερίζεται και η Κομισιόν, ή αν θέλετε, εγώ συμμερίζομαι την εκτίμηση της Κομισιόν. Το σημαντικό ερώτημα τώρα είναι γιατί αυτή η κατάσταση. Γιατί αυτή η κατάφορη άρνηση της Πολωνίας να συμμορφωθεί με τις συστάσεις της Κομισιόν, αλλά και με τις συστάσεις δεκάδων άλλων οργάνων. Δεν υπάρχει όργανο το οποίο να μην έχει αποφανθεί υπέρ αυτή της ανάγκης και που να μην έχει επικρίνει την Πολωνία. Σχετικά με αυτές τις μεταρρυθμίσεις, αν και είναι μεταρρυθμίσεις εντός εισαγωγικών. Λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, αυτό το οποίο έμαθαν οι πολωνικέ αρχές είναι το εξή. Έμαθαν δυστυχώς από την ε, αδράνεια της Ευρωπαϊκή Ένωσης να κάνει κάτι ουσιώδες στην περίπτωση της Ουγγαρίας. Αυτό έμαθαν. Έμαθαν ότι αν κάποιος κολλησιεργήσει αρκετά, προσποιούμενο ότι συμμετέχει στον διάλογο, μπορεί να συνεχίσει να κάνει ό,τι κρίνει σκόπιμο, μέχρι ότου είναι πολύ αργά πια για να ανατραπούν οι επιτοδισμένες αλλαγές. Δυστυχώς η Ευρώπη λοιπόν δίνει ελπίδες στην Πολωνία. Γιατί όλο και περισσότερο όσο περνάει ο χρόνο, θα είναι όλο και πιο δύσκολο να ανατρέψουμε την κατάσταση και να πάμε στην προτεραιά κατάσταση. Κάτι άλλο το οποίο θέλω να πω εδώ είναι το εξή. Μία άλλη όψη του αυταρχισμού της πολωνικής κυβέρνησης είναι η κατάφοροι άγνοια του παράλογου της κατάστασης. Τι εννοώ. Βλέπουμε μια οργουελιανή γλώσσα, μια διπλή γλώσσα η οποία έχει μια τρομακτική διάσταση. Λέει ας πούμε η Πολωνία. Μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης. Υπό το κάλυμα αυτό γίνονται συστηματικές επιθέσεις κατά της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης που είναι βεβαίω στοιχείο κλειδί κάθε δημοκρατίας και της πολωνικής αλλά και προϋπόθεση για να είναι κανεί μέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις εδώ. Όλα αυτά προστατεύονται και προβλέπονται από την συνθήκη. Δεν μπορούν όλα αυτά να είναι στα χέρια ε, ενός ανδρό. Οι δεσμεύσει ω τώρα παραμένουν λοιπόν γράμμα κενό και έχουμε φτάσει το 2018 Ζούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτά τα πράγματα είναι τρομακτικά. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να επενθυμίσω μια άλλη σύσταση την οποία παραβαίνουν συστηματικά οι πολωνικές αρχές και λυπούμε πραγματικά γι' αυτό, αλλά η Κομισιόν έχει κατά επανάληψη ζητήσει οποιασδήποτε αλλαγέ, δεν λέω μεταρρυθμίσει, στο οργανόγραμμα ή και στην οργάνωση γενικότερα τη δικαιοσύνη, να προετοιμάζονται σε στενή συνεργασία με τους δικαστές και όλους τους εμπλεκομένους, όλους τους ενδιαφερμένους. Αυτό δεν έγινε και αυτό θυμίζω ότι είναι η πρώτη σύσταση που διατύπωσε η Κομισιόν το 2016. Το βασικό μου λοιπόν συμπέρασμα είναι το εξή. Το συντομότερο ξυπνήσουμε όλοι εναντί αυτή τη απειλή επιστροφή στο παρελθόν. Το γρηγορότερο θα επανέλθει η συνταγματική τάξη στην Πολωνία. Έτσι θα αποκαταστήσουμε και την καλή, την ομαλή λειτουργία του νόμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην έχετε ψευδεστήσεις. Το πρόβλημα εξαπλώνεται και το διάβαζα σήμερα το πρωί αυτά στο τρένο ερχόμενο στις Βρυξέλλες. Τα ίδια γίνονται στη Ρουμανία. Αυτές οι πρακτικές εξαπλώνονται. Το προηγούμενο πάνελ τα όλα αυτά σε μια συγκριτική βάση, αλλά το διευκρινίζω δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε τη, τη συγκριτική μελέτη του νομού για να βελτιώσουμε την κατάσταση στη χώρα Α, στη χώρα Β. Εδώ γίνεται το αντίθετο. Εδώ τα νομικά συστήματα επιδεινώνονται. Δεν είναι πλέον ανευθυμασια η επίκληση του συγκριτικού δικαίου. Εδώ έχουμε μεταρρυθμίσει που δεν είναι καν συμβατέ με το πρωνικό σύνταγμα. Τι μα νοιάζει τι γίνεται στη Γερμανία. Άρα η συγκριτική μελέτη του δικαίου προκειμένου δεν έχει καμία ε, έννοια, είναι ανεφουσίας. Έχω 10 δευτερόλεπτα. Κάθε πτυχή του κράτους δικαίου, όπως το γνωρίζουμε, απειλείται. Με μήμετρα δεν θα θεραπευθεί η κατάσταση. Δεν γίνεται να γνωρούμε ακόμη τις εξελίξεις. Αν να δράσουμε, πρέπει να δράσουμε σήμερα. Όχι μόνο για την Πολωνία αλλά και για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό τη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πες. Ευχαριστώ πολύ που τηρήσατε το χρόνο σας. Πάμε τώρα στον κύριο Ζήχ, το επόμενο μέλος του πάνελ αυτού. Πρόεδρε, κύριε βουλευτές, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Τα προβλήματα των ε, δικαστικών στην Πολωνία είναι από τα πιο συζητημένα θέματα στην ε, ευρωπαϊκή πολιτική τη σήμερα ημέρα. Έχουν υποθεί πολλά για το θέμα. Αλλά αν κάνετε τι κοιτάξει λεπτομέρειε και αν ε, δει τα επιχειρήματα των μεν και των δε, τότε, τότε μπορεί να διαπιστώσει πώ. τα θέματα είναι πολύ πιο περίπλοκα από όσο φαίνεται με πρώτη ματιά. Ε, βέβαια, γίνεται πάρα πολύ δύσκολο κανεί να κάνει να κάνει μια καταγραφή αυτή τη ε, κατάσταση και να τα εξηγήσει μόνο σε 10 λεπτά, γιατί είναι τόσο περίπλοκα. Τέλο πάντων, σα παραπέμπω στην μελέτη που έχουμε κάνει, σηκώνει το έντυπο ο μιλητής. Ε, ευχαρίστως να σας ε, στείλω αυτή μου τη μελέτη ε, ψηφιακά και για να δούμε τώρα τα βασικότερα σημεία όσον αφορά την κατάσταση της δικαιοσύνης στην Πολωνία και για να κάνουμε τα πράγματα λίγο πιο ενδιαφέροντα θα προσπαθήσω να σας αναπτύξω κάποια επιχειρήματα τα οποία δεν έχετε ακούσει μέχρι τώρα. Πρώτα πρώτα είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι η διαμάχη για τη δικαιοσύνη στην ε, Πολωνία ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2015. Τότε που θεσπίστηκε ένας νόμος όσον αφορά κάποιες αλλαγές από τότε την κυβέρνηση συνασπισμού και είχαμε διάφορες διατάξεις ε, επίμαχες που αφορούσαν την εκλογή και επιλογή των δικαστών που σύμφωνα το Σύνταγμα θα έπρεπε να επιλέγονται και ε, θα πρέπει μάλλον να έχουν επιλεγεί και διοριστεί από το επόμενο κοινοβούλιο. Αυτό κηρύχθηκε αντισταγματικό. Αλλά δεν υπήρξαν ε, φωνές αντίρρησης ούτε από τους ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Πολωνία, ούτε από πουθενά διεθνώς. Άλλα γίνανε μετά που έλαβαν μεγάλη δημοσιότητα. Είναι όλα αυτά τα οποία αναφέρθηκαν στη σημερινή συζήτηση. Όχι, δεν θα κολλήσω σε αυτά. Το επόμενο που πρέπει να σας πω είναι ότι δεν είναι ορθό να λέει ότι σήμερα το συνταγματικό δικαστήριο κατά κάποιο τρόπο είναι υποχείριο της κυβέρνησης. Την περασμένη εβδομάδα το δικαστήριο κήρυξε αντίστοιχα ένα σημαντικό νόμο. Σαφώς κόντρα στις θέσεις της κυβέρνησης. Και υπάρχει μια σειρά αποφάσεων τέτοιων τους τελευταίους μήνες. Ακόμα και σε μια υπόθεση για κάποια κανονιστικά διατάγματα επί των οποίων ο ίδιος ο κύριος ε, Μπόντεναρ είχε συμμετάσχει. Κάπα 17 κάθετος 14. Και έκρινε το δικαστήριο και κάποιες ε, διατάξεις όσον αφορά την ε, έρευνα από αστυνομικού είναι αντισδεγματικές. Αφορούσε έλεγχο αυτοκίνητα και πρόσωπα. Αυτό ήταν βέβαια πολιτικά καυτό γιατί αφορούσε τις διοικητικές αρχές και πολλές φορές ε, είχε ακουστεί αντίθετη φωνή της αντιπολίτευσης. Επομένω όλα αυτά ήταν κατά του Κοινοβουλίου και κατά της κυβέρνησης. Σας παραπέμπω και επίσης στη γνωμοδότηση του κ. Μπόντναρ. Επίσης ήταν ε, η απόφαση ομόφωνη και πρόκειτο για Τέσσερις δικαστές. Οι τέσσερις είχαν διοριστεί τώρα και ο ένας παλιότερα. Παρακαλώ. Η επόμενη φάση της ε, προστριβής για την δικαιοσύνη. Αυτό αφορά την νομοθεσία για τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης στη χώρα. το βασικό πρόβλημα του συστήματος δικαιοσύνης είναι ένα σύστημα που δημιουργεί απουσία εμπιστοσύνη. Και το έχουν πει αυτό πάρα πολύ. Πολλές οι διαφωνίες. Για το πώς ε, ασκείται τη δικαιοσύνη σε επίπεδο ενδίκων μέσων. Ε, βέβαια και είχαμε τρία θεσμικά όργανα τα οποία πέρασαν από αυτή τη μεταρρύθμιση. Πρώτα απ' το ανώτατο δικαστήριο. Δεύτερον, το Εθνικό Δικαστικό Συμβούλιο και όλη η τακτική δικαιοσύνη. Άρα θα πρέπει να σταθούμε σε κάποιες πλευρές της μεταρρύθμισης που δεν έχουν συζητηθεί. Ακόμη γιατί πολλά από τα σημεία προστριβής έχουν ήδη συζητηθεί και να μην τα επαναλαμβάνουμε. Πάντως, πρέπει να αναφέρουμε ότι πολλές μεταρρυθμίσεις πέρασαν χωρίς να ακουστεί αντίθετη φωνή. Και έτσι βελτιώθηκε η διαφάνεια στον τομέα της δικαιοσύνης και η αμεροληψία. Όσον αφορά την κατανομή των υποθέσεων, ας πούμε, στη δικαιοσύνη τώρα, η σύνδεση των δικαστηρίων γίνεται με ε, κομπιούτερ, γίνεται με, τυχαία επιλογή. Και στο στεγματικό δικαστήριο. Η σύνδεση του δικαστήριου γίνεται αλφαβητικά, με βάση τέλο πάντων την αλφάβητα. Ένα παλιότερα δεν μπορούσε να υπάρξει επιρροή επί των αποφάσεων όπως γινόταν δηλαδή ο ορισμός παλαιότερα, γιατί αν υποθέσει υποθέσεις σε συγκεκριμένους δικαστές, πήγαινε σε θα μπορούσαν να μεταφέρονται οι δικαστές από το ένα τμήμα στο άλλο, από το ποινικό, στο πολιτικό κλπ. κλπ. Ε, γι' αυτό σας λέω ότι οι προστριβές αφορούσαν συγκεκριμένες ε, αλλαγές. Ήταν προσωπικά κάποια θέματα που βρήκαν στο επίκεντρο της θύλας. Για να δούμε τώρα κάποια σημαντικά επιχείρηματα. Ο νέος νόμος για το σύστημα λειτουργίας των δικαστηρίων ε, ε, επι... Ε, επικρίθηκε επάφθη ο επικεφαλής του Συμβουλίου των Δικαστών από το Υπουργείο αλλά δεν έγινε κανένα είδου κυνήγημα μαγισσών, κανένα είδου εκαθάριση. Πέρασαν έξι μήνε. 18% των πρόεδρων των δικαστηρίων ε, επάφθησαν, αλλά πια δεν έγινε άλλη τέτοιου είδους ε, απόλυση. Αυτοί πια δεν αναθέτουν ε, υποθέσεις, επομένως δεν έχουν πια τόσο μεγάλη ισχύ στο παρελθόν υπήρχαν τέτοια ζητήματα. Βέβαια, το πιο επίμαχο σημείο είναι αυτό που προβλέπεται και που θεσπίστηκε τον Ιουλίο φέτος για τον το δικαστήριο. Ήδη ακούσαμε μια σειρά επιχειρημάτων για τον νόμο αυτό που διεύρυνε την σύνθεση του δικαστηρίου και ταυτόχρονα κατέβασε το ρίστο εξοδότησης των δικαστών. Ακούσαμε ένα σωρό αμφιβολίες σε σχέση με αυτό. Η, το όριο το οποίο τώρα θεσπίστηκε για τους δικαστές του Αναδότου, είναι 65 για τους άνδρες και 60 για τις γυναίκες. Ε, αυτό δεν διαφέρει από το ότι ισχύει γενικότερα και που σχεδόν ταυτόχρονα θεσπίστηκε. Μετά αυτές τις ε, μεταρρυθμίσεις για τον το δικαστήριο το υποχρεωτικό όριο τώρα εξισώθηκε για γυναίκες και άντρες. Στα 60 πήγε το όριο. Εάν θέλουν μπορούν τότε να αποχωρήσουν. Εδώ είχαμε θέμα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ο εισήγητη του νομοσχεδίου είχε πει ότι βασίζεται η νομική βάση τέλο το άρθρο 180 πρόγραμμα 5 του συντάγματο που μιλάει για του δικαστέ, την πάυση του κλπ. Οι αντίθετοι λένε ότι δεν υπάρχει αναλογία σε τέτοιο μέτρο, ιδίω όσον αφορά για, τον, για την πάυση τέλο πάντων και απόλυση του πρώτου Προέδρου του δικαστήριο. Το ανωτάτο δικαστήριο. Α, θα κλείσουμε δύο πάρα πολύ σύντομα σχόλια. Σας είπα κάποια παραδείγματα για τα θέματα που κατά τη γνώμη μου προέκυψαν στη σημερινή συζήτηση. Ε, βέβαια και πάρα πολλά σημαντικά επιχειρήματα προτάχθηκαν να, τα λάβουμε υπόψη. Απ' την άλλη, ακούστηκαν πάρα πολλές γενικόλογες διατυπώσεις και δηλώσεις. Δεν έλαβαν υπόψη όμως το δικαστικό σώμα θα πρέπει να υπάρχει ένας υποδομητικός διάλογος και να βασίζεται σε στεγανή, σε, σε, σε, σε έγκυρη εξέταση των πραγματικών περιστατικών. Ευχαριστούμε κύριε Λαμψαγγελάρ που προεδρεύσατε για αυτό το τμήμα της συνεδρίας σας. Και ζητώ συγγνώμη και από τον κύριο Πέτς. Και βεβαίως πολύ από το υλικό σας ε, το έχουμε χρησιμοποιήσει και οπωσδήποτε θα απαντήσετε και πολλές ερωτήσεις. Και ξέρω πως πολλοί συναδελφοί σας εργάζεστε πολύ σκληρά στον τομέα αυτόν και το λέω αντικειμενικά αυτό τώρα αν του εάν ε, διαφωνεί ή συμφωνεί κανείς ε, μαζί σας. Λοιπόν, θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Μιχαλοϊκόβιτς, ο οποίος είναι δικηγόρος, ε, θα μας πείτε και εσείς κάποια πράγματα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι. Στην σύντομη παρουσίασή μου θα ήθελα να αναφερθώ ως μαχόμενος δικηγόρος σε κάποιες πρακτικές επιτυχίες της κατάστασης στην Πολωνία που έχουν σχέση με την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Τώρα έχουμε μια κατάσταση όπου έχει γίνει ένα μεγάλο βήμα από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Η καταγγελία της ε, Κομισιόν και τα ενδιάμεσα. Τα προσωρινά μέτρα του ΔΕΚ είναι πολύ σημαντικά μέσα στην μάχη για να σταματήσει η καταστροφή της ανεξάρτητης πολωνικής δικαιοσύνης. Αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση όπου οι δικαστές ε, του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου άνω των 65 ετών έχουν επιστρέψει στην ε, δουλειά τους και δικάζουν. Ο κ. Γκέρσδοφ είναι ο ανώτατος δικαστής μέχρι το 2020. Οπότε η κατάσταση ε, διορθώθηκε από την πλευρά των συνθήκων και την αρχή της αποτελεσματικής δικαστικής ε, προστασίας. Δηλαδή επανήλθε στην κατάσταση 1ης 3ης Απριλίου και του νέου νόμου περί ανώτατου δικαστηρίου. Αναμένουμε λοιπόν τώρα την δίκη και την απόφαση του ΔΕΚ, αλλά αυτό το οποίο θα ήθελα εγώ να τονίσω είναι ότι αυτές οι διαδικασίες μας δείχνουν πόσο σημαντική είναι και πόσο σοβαρό αποτέλεσμα έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί στην Πολωνία τα τελευταία τρία χρόνια όλοι θεωρούσαν ότι τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει αυτόν τον οδοστρωτήρα που κονιορτοποιούσε το δικαστικό μας σύστημα και με τις ε, προσπάθειες ε, του Κοινοβουλίου, της Κομισιόν ε, και του ΔΕΚ που καταφέραμε να σταματήσει αυτό. Γι' αυτό εξ ονόματος της πολιτικής κοινωνίας των πολιτών και της τεράστιας φιλοσοφίας των πολιτών δικηγόρων θα ήθελα από αυτό το βήμα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εσάς και την Κομισιόν για την αποφασιστικότητα και τις προσπάθειες που κάνει την, προσπά... για την προάσπιση του κράτους δικαίου στην Πολωνία. Αλλά η διαδικασία αυτή, η επιπαραβάση που εκκρεμεί τώρα ενώπιν του ΔΕΚ, δυστυχώς δεν αρκεί για να αποκαταστήσει το κράτος δικαίου στην Πολωνία και τα κριτήρια του συστήματος της δικαιοσύνης. Εξακολουθούμε να έχουμε μια συνταγματική κρίση, υπάρχει το σοβαρό πρόβλημα με το συνταγματικό δικαστήριο που έχει παραλύσει και δεν είναι πλέον ανεξάρτητο. Ακούσαμε ήδη αυτά τα οποία μας είπε, τα σύντομα και ουσιαστικά, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής της Βενετίας. Και βεβαίως η έλλειψη ανεξαρτησίας είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα. Αλλά ποιο είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα τώρα. Το προπατορικό αμάρτημα θα έλεγα που δηλητηριάζει ολόκληρο το σύστημα στην Πολωνία είναι το Εθνικό Συμβούλιο Δικαιοσύνης. Επελέγει με έναν τρόπο αντισυνταγματικό που δεν συμβάζεται και με τις διεθνείς προδιαγραφές περί ανεξάρτητης δικαιοσύνης. δεν ε, πλήρει δηλαδή τον συνταγματικό τρόλο. Σύμφωνα με το άρθρο 186 του συντάγματος, το Συμβούλιο δικαιοσύνη θα πρέπει να προστατεύει την ανεξαρτησία των δικαστηρίων και των δικαστών. Εν τω μεταξύ, ε, είναι πλήρως υποτεταγμένο στην ε, εκτελεστική και νομοθετική εξουσία, οπότε πώς μπορεί να διασφαλίσει την ανεξαρτησία της δικαιοσύνη είναι αδύνατον. Και η γνωμοδότηση αυτή επιβεβαιώνεται και από Πολωνούς ε, και ξένους ειδικού του συνταγματικού δικαίου από διεθνείς οργανισμούς. Μας τα είπε και η Κομισιόν, η Επιτροπή της Βενετίας, την οποία επίσης ακούσαμε, το Δίκτυο Συμβουλίων Δικαιοσύνης που επίσης ακούσαμε, το Εθνικό Συμβούλιο Δικαιοσύνης λοιπόν, όπως μας είπε και ο κύριος Στέρκ, η Ευρωπαϊκή Ένωση Συμβουλίων ανέστηλε την συμμετοχή του Πολωνικού Συμβουλίου ακριβώς γιατί δεν θεωρείται ε, πλέον ανεξάρτητο. Αρκεί να δούμε το πώς λειτουργεί στην ε, Πολωνία και το πώς εκφράζονται τα πρόεδρος. Ο πρόεδρος, παραδείγματος χάρη, ο κύριος Μάζουκ, όταν τον ρώτησαν δημοσιογράφοι για το εάν το Εθνικό Συμβούλιο θα σεβαστεί την απόφαση του ΔΕΚ, είπε ότι θα διαβολευτεί με την κυβέρνηση. Γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μια κατάσταση όπου το Εθνικό Συμβούλιο Δικαιοσύνης ε, ανακοίνωσε ότι θα παραπέμψει την υπόθεση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο για να ξεκινήσουν πειθαρχικές διαδικασίες κατά του δικαστού Ζαμπότσκι, του ανωτάτου δικαστηρίου ο οποίος είναι πρόεδρος του ποινικού τμήματος και δεν επέτρεψε σε έναν νέο δικαστή να αναλάβει καθήκοντα γιατί έχει εκλεγεί ε, από το αντισυνταγματικό αυτό συμβούλιο. Γιατί ακριβώς υπάρχει αυτή η προσωρινή διαταγή. Γι' αυτό το έκανε αυτό ο δικαστής ε, Σαμπόσκι. Και για τον λόγο αυτό το νέο Εθνικό Συμβούλιο Δικαιοσύνης τον απειλεί με επιθαρχική διαδικασία. Αυτά έτσι ως ε, παράδειγμα. Ε, να σας πω και άλλο ένα παράδειγμα. Εκπροσωπώ πολλούς δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου άνω των 65 ετών στην έφεση αυτή που υποβάλλουν κατά των αποφάσεων του Εθνικού Συμβουλίου Δικαιοσύνης για αυτούς οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο και το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο. Όταν εγώ και ο συναδελφός μου αποστήλαμε την έφεση απευθείας στο Εθνικό Συμβούλιο Δικαιοσύνης, η απόφαση του Συμβουλίου και θα έπρεπε κανονικά να την μεταβάσει απευθεία στο ανώτατο δικαστήριο, αλλά δεν το έκανε. Χωρί να έχει κάποια αρμοδιότητα, δικονομικά μιλώντα, ε, να εξετάσει την αίτηση αυτή. Αρνήθηκε απλά να την διαβιβάσει στο ανώτατο δικαστήριο. Έτσι λειτουργεί σήμερα το, το Εθνικό Συμβούλιο δικαιοσύνη. και η Δικαστική Ένωση, η Ιουστίτσια, συνέταξε μια ειδική έκθεση για την κατάσταση της δικαιοσύνης με βάση μια ανώνυμη έρευνα των δικαστών. Ε, η Ιουστίτσια έχει 3.000 μέλη δικαστές, σχεδόν το 1 τρίτο των δικαστών και έδειξε ότι το 90% των ερωτήτων θεωρούν ότι το κράτος δικαίου κινδυνεύει. 50% των δικαστών έχουν ήδη δεχτεί πολιτική πίεση. Ε, κάτι το είναι τρομακτικό, καθώς θεωρητικά ζούμε σε μια δημοκρατική χώρα που υποτίθεται ότι σέβεται τις εμελιώδεις αξίες των ευρωπαϊκών συνδικών. 91,5% των δικαστών ε, που ερωτήθηκαν απάντησε ότι το Εθνικό Συμβούλιο Δικαιοσύνη ε, δεν πληρεί τον συνταγματικό του ρόλο και 85% των δικαστών είπαν ότι τα μέλη του Συμβουλίου για Δικαιοσύνη πρέπει να παρατηθούν. Για την πίεση τώρα που υφίστανται οι δικαστές, έχουμε πειθαρχικές διώξεις ε, που στρέφονται κατά των δικαστών εκείνων που μιλούν ε, ρητός για την απειλή που δέχεται το κράτος δικαίου. Και θα λογοδοτήσουν ε, στο πειθαρχικό για το ότι πήγαν στα, μίλησαν στα ΜΜΕ ότι έκαναν εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχολεία ή σε προσωμιώσεις δίκης. Ένα καλό σχόλιο για αυτό το οποίο είπε ο κύριος Σκάρσκι περί πολιτικών υποτίθεται δραστηριοτήτων των δικαστών. Δηλαδή ακούγεται απίστευτο, αλλά ε, δυστυχώς είναι η αλήθεια. Ένα πρόγραμμα το οποίο λέγεται Συνταγματική Εβδομάδα, που οργάνωσε μια ΜΚΟ του καθηγητή Χάουντα που λαμβάνει ε, χώρα κάθε χρόνο σε πολλά σχολεία και συμμετέχουν γύρω στους 600 δικηγόρους σε αυτό και το κάνουν δωρεάν. Δικαστές, ε, εισαγγελείς, δικηγόροι και κάθε φορά απευθύνεται σε 50.000 παιδιά και ε, πολλές φορές ε, τον προηγούμενο βήμα Υπάρχουν προσπαθίε για να εκφοβιστούν αυτοί οι δικηγόροι και οι δικαστές και οι εισαγγελίε. Ναι, ναι, ολοκληρώνω. Λοιπόν, θα ήθελα όμως να τονίσω ότι οι Πολωνοί δικαστές ε, αντιστέκονται γενναία και παραμένουν ανεξάρτητοι παρά το ότι αυτό βεβαίω έχει ένα χαρακτήρα ο οποίος ίσως ε, του κάνει να το σκεφτούν ε, να το ξανασκεφτούν πριν κάνει κάτι. Λοιπόν, έχουμε αυτή την Επιτροπή για την Υπεράσπιση τη δικαιοσύνη από 12 οργανώσει, Διεθνή Αμνηστία, το Ίδρυμα του Ελσίνκη, Ενώσεις Δικαστών κτλ. Άρα έχουμε νομική στήριξη και ηθική στήριξη σε όλους τους διοκόμενους δικαστές και παρακολουθούμε όλες τις περιπτώσεις διώξεων κατά δικαστών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ και για τη βοήθειά σας όταν σας επισκεφθήκαμε. Ευχαριστούμε την Free Courts. Και τώρα, κυρία Σουλέκα, από το Ίδρυμα Στολσίνκη για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Κυρίε και κύριοι, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την ευκαιρία να πω δύο λόγια εκ μέρου του Ιδρύματο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου του Ελσίνκη για την κατάσταση στην Πολωνία. το Ίδρυμά μας. Έχει ενδική παρουσία στην Πολωνία, εδώ και 30 χρόνια θα έλεγα. Παρακολουθούμε την κατάσταση και περιμενόμεθα υποθέσεων δικαιωμάτων του ανθρώπου. Τον Ιούνιο του 2015, μάλιστα, διαμαρτυρηθήκαμε και για τις αλλαγές στο συνταγματικό δικαστήριο. το 2015 στην Πολωνία γινόμαστε μάρτυρες ε, προσπαθειών άνευ να πληγεί η δημοκρατία. Οι αλλαγέ αφορούν σχεδόν κάθε πτύχη της δημοκρατίας, αφορούν τη δικαιοσύνη, τα μέσα, την ελευθερία των μέσων και την λειτουργία των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Από συστημικής απόψεως, Καμία από αυτέ τι αλλαγέ δεν αποτελεί απαραίτητη μεταρρύθμιση. Δεν πρόκειται για μεταρρυθμίσει βεβαίω. Πρόκειται για απόπειρε να υπονομεύσουν την ανεξαρτησία όλων αυτών των φορέων. Οι αλλαγέ είναι πρώτον νομοθετικέ. Αποσκοπούν στο να παραλύσουν κάποιου θεσμού και να του εξαρτήσουν από την πολιτική εξουσία. Συνοδεύεται πολλές φορές από πολιτικές αλλαγές, τροποποιήσεις για να καταπνιγούν οι οργανισμοί αυτοί στη λειτουργία τους. Το πιο ανησυχητικό είναι όμως ότι υπάρχει μια εχθρική ατμόσφαιρα, υπάρχει στοχοποίηση συγκεκριμένων ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και συγκεκριμένων δικαστών, εισαγγελέων και μέσων. Οι αλλαγές αυτές διακρίνονται επίσης η ε, την ακόρεστη ε, πίνα, θα έλεγα, της κυβέρνηση να διορίζει τους πάντες και τα πάντα παντού. Δύο παραδείγματα τα οποία αποδεικνύουν τη φύση αυτών των αλλαγών είναι τα εξή. Πρώτον, η δικαιοσύνη. Βέβαια, μετά από τα όσα ακούσατε, ε, νομίζω θα πλήξταν ξανά από τι συμβαίνει στην δικαιοσύνη, αλλά αξίζει τον κόπο. Δώστε μου δύο λεπτά. 15 νομοθετήματα που διέπουν την δικαιοσύνη ψηφίστηκαν από την κυβερνητική πλειοψηφία. Κανένας όμως από αυτούς τους νόμους, τους 15 νόμους, δεν ε, αποσκοπεί στην επίλυση κάποιου ζωτικού προβλήματος. Ε, για παράδειγμα, η ερχοπορία της δικαιοσύνης, η διευκόλυνση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη ανθρώπων με αναπηρίες, αύξηση του προσωπικού κλπ. Αντιθέτως, όλες οι αλλαγές αποσκοπούν στο να καταργήσουν κάθε ανεξαρτησία των δικαστών οι διορισμοί από εδώ και πέρα θα είναι καθαρά πολιτικοί. Οι συνδελφοί μου και εγώ, αλλά και τα μέλη του προηγούμενου πάνελ, μίλησαν για ανώτερο Συμβούλιο Δικαιοσύνη, για ανώτερο Δικαστήριο, το Συνταγματικό Δικαστήριο και ούτω καθεξής. Αλλά εγώ θέλω να πω δύο λόγια για τα όσα το 2017 και 2018. Οπότε η δικαιοσύνη πέρασε διαπηρώσει και σιδήρου, ξεκινώντας από την απόλυση του Πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών. Να σου πω μάλιστα ότι πρόκειται για έναν δικαστή επί τρία ο που ήταν πρόεδρος του Ανατολικού Δικαστηρίου τα τελευταία 8 χρόνια και ο οποίος αποπέμφθηκε με απόφαση μια γραμμή που του εστάλει από το Υπουργείο Δικαιοσύνη με φάξ, παρακαλώ. Άλλαξαν επίση οι πρόεδροι των δικαστηριών και με τρόπο μυστικό. Ένα συγκεκριμένο δικαστή έμαθε για την προσπάθεια να εκπαραθυρωθεί επειδή δεν έβγαλε αποφάσεις που άρεσαν στην κυβέρνηση. Κάποιοι μάλιστα επιβουλεύτηκαν την θέση του και έτσι κάπως έμαθε την προσπάθεια της κυβέρνησης. Επίσης, ο διορισμό του νέου δικαστή έγινε χωρίς την σύμφωνη γνώμη των άλλων δικαστών. Και το ακόμα πιο ανησυχητικό είναι ότι οι νέοι επικεφαλεί δικαστές είναι δικαστές οι οποίοι υπό κανονικέ συνθήκε σε καμία περίπτωση δεν θα είχαν ε, λόγω απειρία την δυνατότητα να καταλάβουν θέσει επικεφαλής δικαστηρίων. Να επιστήσω επίσης την προσοχή σας σε ένα άλλο ζήτημα. Η κρίση του κρατούς δικαίου, τη οποία γινόμαστε μάρτυρες τα τελευταία τρία χρόνια, έχει αντίκτυπο σε κάθε πτυχή της λειτουργίας του κράτους και των ανεξαρτήτων αρχών και θεσμών. Κάτι το οποίο ξεχάσαμε στη συζήτηση αυτή. Τα τελευταία τρία χρόνια η Πολωνική Ομοσπονδία ΜΚΟ κατέγραψε δεκάδες παραδείγματα παράβασης των κανόνων και της ελευθερίας συνεργασίας μεταξύ των ΜΚΟ. Επίσης παρατηρούμε παραδείγματα περάτωσης της συνεργασίας ΜΚΟ με την δημοσία διοίκηση και συστημική προτιμησιακή πολιτική στη διανομή των δημοσίων κονδυλίων. αυτά δεν συνάδουν με την δικαιωμένη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ της κοινωνίας των πολιτών. Κάποιες ε, ΜΚΟ αποκοπτώνται από τα έσοδά τους, ειδικά αυτέ που υπερμείνονται των δικαιωμάτων των γυναικών, μειονοτήτων κλπ. Πολλέ φορέ δέχονται υποθέσει ή αποκόπτονται, απορρίπτονται από την διαδικασία δημόσια διαβούλευση. Στην Πολωνία τα τελευταία τρία χρόνια τα πιο βασικά νομοθετήματα, αυτά τα οποία είναι τα πιο σημαντικά δηλαδή από συστημικής απόψεως, ψηφίστηκαν με συνοπτικές διαδικασίες χωρίς διαβούλευση. Οι επιθέσεις όμως κατά του κρατούς δικαίου δεν είναι μόνο αυτές. Πρέπει η διεθνή κοινότητα να συνεχίσει να παρακολουθεί την κατάσταση από κοντά για να θέσει τέλος στην απειλή αυτή επειδή έχω τρία λεπτά ακόμη, ε, επιτρέψτε μου να σταματήσω και να αφήσω αυτά τα τρία λεπτά για ερωτήσει και απαντήσεις. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ναι, 7 λεπτά όντως, ναι, ναι, τα κατάφερες 7 λεπτά. Ναι, δεν μετράει η ποσότητα, αλλά η ποιότητα. Ελπίζω να μπορέσω να το πω αυτό και στο τέλος. Σαν χαϊκού ακούστηκε. Τέλεια. Τα είπατε μια χαρά. Και να πω και προς τους αδέλφους μου, αν και καθυστέρησε λίγο. έχει το ρόλο σας ως ακτιβίστρια. Ξέρω ότι παρεμβαίνετε όλοι σας σε ένα φορτισμένο περιβάλλον, ε, αλλά έχουν πολύ μεγάλη σημασία όλα αυτά για την κοινωνία των πολιτών και για τις οργανώσεις της. Ως πανεπιστημιακή έχετε πολύ σημαντικό ρόλο λοιπόν και σας ευχαριστώ γι' αυτό που μας ενημερώνετε για την κατάσταση. Σας ευχαριστώ πραγματικά πολύ. Και να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους, τους βουλευτές που παραμένουν στην αίθουσα, ήταν αρκετά μακροσκελής και παραμένει μακροσκελής η ακρόαση, η Μπάρμπαρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, επίτρεψέ μου να διαφωνήσω με αυτό το τελευταίο που είπες. Ότι δηλαδή όλα όσα ακούσαμε ήταν συγκεκριμένα, ισορροπημένα. Εγώ έχω πάντως ένα ερώτημα που ακριβώς αυτό αφορά. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Ζήχ. Ήταν επιστημονικά το όσα μας είπατε κύριε Ζήχ και το άρθρο σας η νομική δεν έχει αποχρώσεις εθνικιστικές και προηγουμένως ο καθηγητής, ο κύριος Σάουσεν μας μίλησε για διαφορετικές ε, νομικές παραδόσεις Μισό λεπτό, δεν τέλειωσα, δεν τέλειωσα την ερώτησή μου. Επομένως η νομική έχει έναν ε, παγκόσμιο χαρακτήρα κατά κάποιο τρόπο. Όταν γράφετε άρθρα έχετε επιστημονική μεθοδολογία και όταν ε, παρουσιάσετε τις ε, απόψεις, γιατί αυτές οι μισές αλήθειες, αυτά τα περίεργα επιχειρήματα που εκτίθενται. Να, ας πούμε, μιλήσατε για αυτή την πλατφόρμα το 2015 για τους διορισμούς των ε, δικαστών στο Δημοτικό Δικαστήριο αλλά την ίδια χρονιά το Δημοτικό Δικαστήριο απεφάνθη και έκρινε σαφώς ότι δύο διοριστέντες δικαστές από το προηγουμένο Κοινοβουλίου ε, διορίστηκαν με τρόπο αντισταγματικό. Να τι θα πει ε, νόμος. Α, και ανετράπει τέλο πάντων το ε, διάταγμα που τους διόρισε. Την επόμενη φορά που θα κάνετε μια ομιλία, αν αρχίσετε από το 2015, παρακαλώ, και αυτό να αναφέρετε. επρόκειτο για μέλη της πλατφόρμας που προσέφυγαν. Τώρα κάτι άλλο. Τι γίνεται με την τυχαία επιλογή των δικαστών που θα διορίζονται. Αυτό ξεκίνησε πρώτα-πρώτα τον Δεκέμβριο του 10. Ε, ναι, μάλλον θα ξεκινήσει, συγγνώμη. Ακόμα δεν έχει χρησιμοποιηθεί αυτή η μέθοδος. Και σας ε, παραπέμπω στην ε, Ζεποτσπόρτα, την εφημερίδα. Εκεί υπάρχει ένα άρθρο λοιπόν το οποίο κατά αναφέρει το πώς γίνεται η ηλεκτρονική επιλογή ε, των ε, δικαστών και ηλεκτρονικά του αντίθενται δηλαδή οι υποθέσεις. Στο παρελθόν υπήρχε ηλεκτρονική επιλογή. Το ποιο δηλαδή θα δικάσει ποια υπόθεση. Τώρα, όσον αφορά το όριο συνταξιοδότησης, δεν θέλω να διαφωνήσουμε. Αλλά στο δικαστήριο και στο Ισλαμικό δικαστήριο όλοι οι δικαστές υποστηρίζουν ας πούμε το ΠΙΣ, εάν όλοι μάλλον ε, υποστήριζαν το κυβερνητικό κόμμα το ΠΙΣ, τότε θα τους ε, διορίζαμε για όλη τους τη ζωή. Γι' αυτό σας παρακαλώ πέστε μου εσείς όταν κάνετε μια ανάλυση αναφέρεστε στις διαφορετικές απόψεις κάποιων διεθνών οργανισμών. Φιλτράρετε έτσι τα επιχειρήματά σας. Πάρα πολύ σύντομα θα απαντήσω. Μισό λεπτό λέει ο πρόεδρος, μισό λεπτό. Γιατί υπάρχει και πρόεδρος στην αίθουσα. Η Μπάρμπαρα Σπινέλη έχει το λόγο. Όχι, όχι, αποσύρω. Γιατί έχει πάει εξι ώρα. Θα φύγουν, θα φύγουν οι διερμήνες. Άρα μας τα πείτε στα αγγλικά. I, I'm very happy to uh, hear this uh, question. Uh, να, να σας ε, απαντήσω κύριε Κοντρίτσικα, προς έκπληξή σας. Θα συμφωνήσω με τα περισσότερα από όσα είπατε. Αυτά όλα τα πραγματικά περιστατικά που μας ε, αναφέρατε. Διαβάστε προσεκτικά τα άρθρα μου, αυτά που αναφερθήκατε. Ε, εκεί θα δείτε ότι αποτυπώνω όλα αυτά. Όπως όμως είπα αρχή-αρχή στην ε, δεκάλεπτη ζήγησή μου, προσπάθησα να αναφερθώ στα όσα δεν είχαν αναφερθεί στη σημερινή συζήτηση. Δηλαδή είπα πράγματα που κανείς άλλος δεν τα είχε αναφέρει. Um, well, that was an interesting answer. <laughs> Πολύ ενδιαφέρουσα η απάντησή σας. Όχι, όχι, απλώς προσπάθησα αυτό, να, να, να πω αυτά που δεν είπαν οι άλλοι, τα κενά που είχαν αφήσει, να τα... Ε, Άρα, δεν έκανα μια πολιτική ομιλία. Μπάρμπαρα. εκπροσωπείται ένα πάρα πολύ αξιόλογο πανεπιστήμιο. Καθολικό. Δεν είναι κανένα περιφερειακό, επαρχιακό δικαστήριο. Αυτά περίμενα από σας, τα καλύτερα. Όχι, δεν είναι ιδιωτικό, δεν είναι ιδιωτικό. Καλά, καλά. Θα τα πούμε και άλλο αν θέλετε. είχαμε ερωτήσει προ όλου, αλλά να του ευχαριστήσουμε όλου, όχι μόνο για όσα είπαν σήμερα, αλλά και για όλα όσα έκαναν για να μα βοηθήσουν όταν κάναμε την αποστολή. Ε, γιατί δεν είναι μόνο τόσο όσα κάνετε σήμερα, είναι τα όσα ε, κάνετε ως προετοιμασία και όσα θα συνεχίσετε να κάνετε. Τώρα θα φύγουν οι διερμηνείς ε, συνάδελφοι. Οπότε θέλω να ευχαριστήσω του όσους συναδέλφους ε, ήρθαν. Χουαν Φεράντο, η Μπάρμπαρα, η άλλη Μπάρμπαρα, ο Μίχαλ μόλις έφυγε. Ευχαριστώ όλους για τους συνεργάτες μας. Καλά είχα πολλά να πω για να κλείσω την ακρόαση, αλλά τέλος πάντων έχω στείλει το σχέδιο της έκτης πολιτικής ομάδας. Ε, κάποιοι συναδελφοί έχουν δει το σχέδιο κειμένου τα στείλαμε και στην μόνιμη αντιπροσωπεία της Πολωνίας Άρα η κυβέρνηση θα λάβει γνώση, έντος εβδομάδας μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις και είπαμε ότι θα δημοσιοποιηθεί τον ε, Δεκέμβριο το κείμενο. Δεν υπάρχει πολλής χρόνος μέχρι τότε. Άρα θα ολοκληρώσουμε τη διαδικασία μας. Και συγγνώμη για τους αδέλφους που είναι εδώ και δεν ξέρω το όνοματά τους και τους ευχαρίστησε. Άρα θα είμαστε σε επαφή. Ευχαριστούμε το χρόνο σας, προσπαθειές σας. Μπράβο που αντέξατε σήμερα. Αν τα ξαναπούμε τον Δεκέμβριο που θα έχουμε το σχέδιο κειμένου και θα συνεχίσουμε τότε.